Αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε στο δεύτερο μέρος της συνεδρίασής μας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Και θέλω ιδιαίτερα θερμά να καλωσορίσω εδώ τον Ισπανό Υφυπουργό Αρμόδιο για θέματα Ευρωπαϊκή Ένωση, τον κύριο Τιέγκο Λόμπε Γαρίδο, ο οποίο συχνά έρχεται εδώ στην Επιτροπή μα, κάτι το οποίο μα χαροποιεί όλο ιδιαίτερω. Είναι πολύ καλές οι σχέσεις που έχουμε με την Ισπανική Προεδρία. Το ότι έρχεστε εδώ στην Επιτροπή μας και το ότι καλείτε και τους συναδέρφους να έρχονται και να συμμετέχουν σε διασκέψεις, σεμινάρια κλπ. Είναι πάρα πολύ θετικό. Κύριε Βανιού, για παράδειγμα, πρόσφατα προσκαλέθηκε στην Πάλμα Ντε Μαγιόρκα για τα θέματα καταναλωτών, δικαιώματα καταναλωτών. Πολύ καλό αυτό. Επίσης θέλω εδώ εκ μέρους όλων να σας ευχαριστήσω που με προσκαλέσατε στο γεύμα που είχατε με το Συμβούλιο Ανταγωνισμού τον Μάιο στις Βρυξέλλες, όπου και μπορέσαμε να συζητήσουμε λιγάκι για τη δουλειά μας όσον αφορά την εσωτερική αγορά. Ήταν πολύ χρήσιμο, πιστεύω. Μας ε, βοήθησε να μιλήσουμε και για την έκθεση του κύριου Μόντι. Πράγματα όπως είπα, χρήσιμα για μας και γι' αυτό ήθελα να το αναφέρω. Λοιπόν, τώρα θα ζητήσω από τον Υφυπουργό να πάρει το λόγο και στη συνέχεια θα ακούσουμε ερωτήσεις. Έχετε μία ώρα στη διάθεσή σας από ό,τι έχω καταλάβει, μετά παίρνετε το αεροπλάνο για τη Μαδρίτη. Οπότε, μία ώρα να μας παρουσιάσετε την ε, προεδρία σας που ολοκληρώνεται και μετά να συζητήσουμε τι μένει ακόμα να γίνει. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Είμαι και εγώ πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ μαζί σας στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όντως, το Μάρτιο ήμουν πάλι εδώ, όπου παρουσίασα τις προτεραιότητες τότε της Ισπανικής κυβέρνησης σε θέματα εσωτερικής αγοράς για το εξάμεινο της Προεδρίας μας. Είμαι εδώ υπό την ιδιότητα του υπεύθυνου, το εξάμεινο αυτό, της Προεδρίας του Συμβουλίου για θέματα ανταγωνιστικότητας στον τομέα που έχει να κάνει με την εσωτερική αγορά. Συνεπώς θα ήθελα να σας μιλήσω εδώ για το τι κάναμε εμείς αυτούς τους τελευταίους μήνες στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας, τμήμα Εσωτερική Αγορά. Τα θέματα θα σας πω στα οποία πετύχαμε συμφωνία, πού προχωρήσαμε, πού μείναμε πίσω τι έχει μείνει δηλαδή για την επόμενη Προεδρία, την Βελγική, η οποία μαζί με την Ισπανία και μαζί με την Ουγγαρία αποτελούν ε, την τριάδα των Προεδριών. Που σημαίνει ότι συνεργαζόμαστε. Υπάρχουν δηλαδή πράγματα τα οποία ξεκίνησαν υπό Ισπανική Προεδρία και θα συνεχιστούν υπό Βελγική Προεδρία. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από το πρόγραμμα της Τριάδας των Προεδριών που ενέκρινε το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων ομόφωνα πριν από έξι μήνες. Τώρα, θα ήθελα να χωρίσω την παρουσίασή μου σε δύο τμήματα. Το πρώτο έχει να κάνει με το νέο ξεκίνημα της εσωτερικής αγοράς. Νομίζω ότι είναι ένα από τα στρατηγικά σημεία, από τα πιο σημαντικά στοιχεία για το παρόν και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρα και για την Ισπανική Προεδρία του Συμβουλίου. Είναι κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολύ τη δικιά σας Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως επίσης ενδιαφέρει ιδιαίτερα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το δεύτερο τμήμα της παρουσίασής μου θα είναι πρωτοβουλίες, θέματα πιο συγκεκριμένα, που υπήρξαν στην ημερήσια διάταξη του τελευταίου αυτού εξαμήνου για μας. Τόσο το Συμβούλιο, όσο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δούλεψαν προκειμένου, μια που είμαστε τα δύο όργανα που συνομοθετούν, προκειμένου λοιπόν μετά από πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προχωρήσουμε στην εκπόνηση νομοθεσίας. Ξεκινάμε το πρώτο τμήμα, με τα οριζόντια θέματα δηλαδή που έχουν να κάνουν με το νέο ξεκίνημα της εσωτερικής αγοράς, τη νέα όθηση. Ήταν ε, κεντρικό σημείο κατά τη διάρκεια της Ισπανικής Προεδρίας του Συμβουλίου. Στις διάφορες συνεδριάσεις που είχαμε στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας, εσωτερική αγορά, το θέμα αυτό είχε κεντρικό ρόλο κεντρική θέση. Πάνω απ' όλα χρειάζεται οικονομική ανάκαμψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και περισσότερο από ποτέ σήμερα η εσωτερική αγορά μπορεί να προσφέρει για αυτήν την οικονομική ανάκαμψη. Μια οικονομική ανάκαμψη διώσιμη. Πριν από μερικές μέρες, μάλιστα, σε μια τελευταία συνάντηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σήμερα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξέρω ότι συζητούν τα μέλη με τον Herman Van Rompuy. Ε, λοιπόν, σε αυτήν ε, τη συνάντηση που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα υπήρξε μνήα στα συμπεράσματα στην Ευρωπαϊκή Ενία Αγορά. Δηλαδή, περνάμε από το ποιοτικό άλμα σε ένα άλλο στάδιο που είναι νέα όθηση με διάφορες πρωτοβουλίες οι οποίες πάρα πολύ καλά συμπεριλαμβάνονται στην πρόσφατη έκθεση του καθηγητή Μάριο Μόντι για μια νέα στρατηγική σχετική με την ενιαία αγορά. Μάλιστα έχω το κείμενο εδώ μπροστά μου. Κείμενο το οποίο επιβλήθη στον πρόεδρο Μπαρόσο στις 9 Μαΐου του 2010. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να υποβάλει προτάσεις προκειμένου να προχωρήσουμε περισσότερο προς την κατεύθυνση της έκθεσης Μόντι και αυτό θα γίνει το φθινόπωρο. Το Συμβούλιο το Δεκέμβριο θα πρέπει να επανέλθει σε αυτό το θέμα. Συνεπώς, η εσωτερική αγορά αποτελεί ένα από τα σημεία στρατηγικής σημασίας για την Ευρώπη του 2020 με στρατηγική, με οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση. Με την πρωτοβουλία λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ζήτησε την έκθεση από τον Μάριο Μόντι και με την πρωτοβουλία του Συμβουλίου, το οποίο προέδρευε η Ισπανία το τελευταίο εξάμεινο και με την πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επίσης που συμμετείχε, στην πρωτοβουλία αυτή και στον προβληματισμό αυτό πιστεύω ότι προχωρήσαμε πολύ. Όπως γνωρίζετε, το Συμβούλιο ανταγωνιστικότητα τις δύο φορές που συνεδρίασε το εξάμεινο αυτό ζήτησε από τον καθηγητή Μόντι να εξηγήσει Καταρχήν τον προσκάλεσαν πριν βέβαια τελειώσει η έκθεση και όταν για δεύτερη φορά είχε τελειώσει η έκθεση, όπου μάλιστα ήταν και ο πρόεδρος της Επιτροπής αυτής, ε, είχατε προσκληθεί κι εσείς τότε. Ήταν τη μέρα που είχα έρθει εγώ εδώ. Και που μάλιστα είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις και σαν τυπογεύμα με όλους τους υπουργούς που ασχολούνται με την ανταγωνιστικότητα στην εσωτερική αγορά. Θα θυμόσαστε πάρα πολύ καλά εκείνη την ημέρα γιατί η συνάντηση αυτή που είχαμε με τον καθηγητή Μόντι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Εμείς λοιπόν κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας τι κάναμε. Συνεχίσαμε με συνεδριάσεις. Είχαμε ξεκινήσει κάπως και κατά τη διάρκεια της Σουηδικής Προεδρίας, αλλά σιγά σιγά προχωρήσαμε και ο καθηγητής Μόντι φροντίσαμε να συμμετέχει στις συζητήσεις μας γιατί πιστεύουμε ότι η έκθεσή του αυτή θα αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς πολύ σημαντικό για τις μελλοντικέ εργασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να δοθεί νέα όθηση στην εσωτερική αγορά. Γνωρίζετε και ο πρόεδρος Μάλκομ Χάρμπορ και εσείς όλοι γνωρίζετε λοιπόν πολύ καλά ότι η εσωτερική αγορά η εμβάθυνσή της είναι ένα σημείο κεντρικής σημασίας, ζωτικής σημασίας, κεντρικό. Είναι κάτι πολύ βασικό που προσέφερε η Ισπανική Προεδρία αυτό το εξάμεινο. Στη συνάντηση εκείνη θέλω να θυμίσω και στην πρώτη συνάντηση με τον Μάριο Μόντι αλλά και στη δεύτερη στο γεύμα όπου ήταν και ο Μάλκορ Χάρμπορ πρόεδρος της Επιτροπής αυτής ήταν παρόν και ο Αντιπρόεδρος Ταγιάννη και ο Επίτροπος Μπαρνιέ που έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην εξέλιξη των θεμάτων αυτών. Στη συζήτηση που έγινε φάνηκε ο ρόλος που πρέπει να παίξει η εσωτερική αγορά ιδιαίτερα μάλιστα στο σημερινό πλαίσιο οικονομικής κρίσης. Η εσωτερική αγορά αποτελεί ένα σημαντικό μέσο προκειμένου να βγούμε από την κρίση, γιατί βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα, ευνοεί την ε, ανάπτυξη και καταργεί εμπόδια και φραγμούς στο εμπόριο. Άρα, συνεισφέρει με αποφασιστική σημασία στην οικονομική ανάπτυξη που αποτελεί και τον κύριο στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κύριο στόχο συνεπώς και της εξάμηνης Ισπανικής Προεδρίας. Έλεγα και θέλω να το υπενθυμίσω πάλι εκείνο το γεύμα που είχαμε με τον καθηγητή Μόντι, τότε λέγαμε με τον Επίτροπο Παρνιέ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια πλήρης εφαρμογή των διατάξεων για την εσωτερική αγορά, για παράδειγμα δική για τι υπηρεσίε θα αναφερθώ σε αυτήν μετά, σημαίνει για την Ευρωπαϊκή Ένωση σημαντική αύξηση του ε, καθάριστου εγχώριου προϊόντος, αλλά και αύξηση της απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα μάλιστα που ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση. Αναφέρθηκε ο Επίτροπος Μπαρνιέ και στην Οδηγία για τις Υπηρεσίες και θα σας μιλήσω για αυτήν και εγώ αργότερα. Ο προβληματισμός των τελευταίων αυτών μηνών και οικονομικά και πολιτικά στρατηγικής σημασίας, ο προβληματισμός αυτός λοιπόν μας οδηγεί στο εξής. Κάποια μέτρα τομεακά, ανακλάδο, δεν φτάνουν προκειμένου να ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά. Άρα χρειάζεται ακόμα πρόοδο σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο για να ξεπεράσουμε τις αντιστάσεις που υπάρχουν. Τους στραγγαλισμούς που θα έλεγα ότι υπάρχουν μερικές φορές στην εσωτερική αγορά, τα διέξοδα τα οποία πρέπει να ξεπεράσουμε. Αυτό θα το πετύχουμε με συνοδευτικές πολιτικές. Για παράδειγμα, βιομηχανική πολιτική, φορολογικό συντονισμός, πολιτική υπέρ του περιβάλλοντος. Και όλα αυτά για να μπορέσουμε να βαθύνουμε περισσότερο στην εσωτερική αγορά. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε βέβαια και την εξωτερική διάσταση της εσωτερικής αγοράς, ούτε τη σημασία που έχουν συγκεκριμένες πτυχές. Αναφέρθηκα πριν στις υπηρεσίες. Υπάρχει όμως και η ψηφιακή Ευρώπη. Μην ξεχνάμε ότι μόλις εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μάλλον από το Συμβούλιο μετά από πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η λεγόμενη Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Ατζέντα, που, στήριξε στις 17 Ιουνίου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι μια από τις πρώτες πρωτοβουλίες, το Flagship Initiatives, που θα είναι μια σειρά πρωτοβουλειών που θα αναλάβουμε φέτος, επτά συγκεκριμένες πολιτικές που εκφράζουν στην πράξη πολύ συγκεκριμένα και που περιλαμβάνονται στη στρατηγική του 2020. Θέλω λοιπόν να αναφερθώ και στην έκθεση Μόντι, αλλά και σε διάφορες ιδέες που ξεκίνησαν από εδώ, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εώθηση στην εσωτερική αγορά. Έκθεση, για παράδειγμα, του Λουίς Γκρέχ για το πώς μπορούμε να προσφέρουμε την εσωτερική αγορά στους καταναλωτές και στους πολίτες. Δηλαδή, δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στον Ευρωπαίο καταναλωτή ο οποίος πρέπει να καταλάβει ότι η ενιαία αγορά είναι μια παραπάνω αξία για αυτόν, ότι βελτιώνει την καθημερινή του ζωή. Υπενθυμίζω, μάλιστα, ότι αυτό ήταν και ένα από τα βασικά στοιχεία της Ισπανικής Προεδρίας, δηλαδή η προσέγγιση στον πολίτη, πώς δηλαδή θα βελτιώσουμε την καθημερινότητα του Ευρωπαίου πολίτη. Υπάρχει επίσης και έκθεση Λαμασούρ για τον ε, πολίτη και τα δικαιώματά του από το 2008 που έχει άμεσα να κάνει με την εσωτερική ενιαία αγορά. Προς αυτή την κατεύθυνση έδρασαν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και το Συμβούλιο το τελευταίο εξάμεινο υπό Ισπανική Προεδρία. Πολύ γρήγορα τώρα θα αναφερθώ λιγάκι σε συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία αποτέλεσαν ε, αντικείμενο των εργασιών του Συμβουλίου, της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βεβαίως. Γρήγορα θα σας τα πω, για να μπορέσουμε, εφόσον το επιθυμείτε, να εμβαθύνουμε περισσότερο σε μερικά από αυτά, εφόσον το ζητήσετε. Ξεκινάω λοιπόν με την οδηγία για τις υπηρεσίες, την οποία αναφέρθηκα πριν από λίγο. Η οδηγία για τις υπηρεσίες σημαίνει οδηγία για ένα τομέα της ευρωπαϊκής οικονομίας που είναι γύρω στο 60-65% του ΕΠ. Και σίγουρα είναι πάνω από 60% όσον αφορά τις θέσεις απασχόλησης. Ζωτική σημασία λοιπόν ο τομέας αυτός. Υπήρξαν εσωτερικές δυσκολίες, αδιέξοδα, σε εσωτερικό επίπεδο, τα οποία εμπόδισαν την ανάπτυξη της αγοράς αυτής υπηρεσιών, που θα βοηθούσε ακόμα περισσότερο στην ανάπτυξη και σε θέσεις απασχόλησης ποιότητας. Πρόκειται για μια από τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, τις πιο μεγάλες που είχε ποτέ στην ιστορία της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα που μιλάμε για τη στρατηγική του 2020 και για το ότι χρειάζονται διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ε, λοιπόν η οδηγία για τις υπηρεσίε αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μένει βέβαια να ενσωματωθεί πλήρω στην νομοθεσία των κρατών μελών. Η προθεσμία έληξε πέρυσι, αλλά ορισμένες χώρες μέλη δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει στην νομοθεσία τους την οδηγία αυτή. Στη συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητα που έλαβαν χώρα το εξάμεινο αυτό, δώσαμε μεγάλη σημασία στο θέμα της μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των χωρών μελών τη οδηγία για τις υπηρεσίες. Είμαστε σε ένα σημαντικό στάδιο αμοιβαία αξιολόγηση. Αφιερώθηκε σε αυτό το θέμα και το τελευταίο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητα. Η άσκηση αυτή λοιπόν τη αμοιβαία αξιολόγηση είναι κάτι που θα κρατήσει όλη τη χρονιά και για μα είναι ζωτική σημασία προκειμένου οι καλέ πρακτικέ των χωρών ε, μελών να γίνουν γνωστέ και έτσι να μπορέσει να εφαρμοστεί πραγματικά στην πράξη Πλήρω η οδηγία για τις υπηρεσίες. Ελπίζουμε το Δεκέμβριο να έχουμε έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, έτσι όπως προβλέπεται από το άρθρο 30 της οδηγίας. Υπάρχει και μια άλλη οδηγία, πολύ σημαντική, ιδιαίτερα σήμερα που είμαστε σε περίοδο κρίσης και μάλιστα σημαντική ιδιαίτερα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Είναι η οδηγία καταπολέμησης των καθυστερημένων πληρωμών σε, στο θέμα του εμπορίου. Ορισμένες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Και το θέμα της οικονομικής κρίσης, η οικονομική κρίση δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την κατάστασή τους. Υπάρχουν δυσκολίες επίσης πρόσβασης σε πιστώσεις. Τις αντιμετωπίζουν πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Οπότε έχει μεγάλη σημασία να ε, εμβαθύνουμε στο θέμα αυτό. Οι καθυστερήσεις πληρωμών οδηγούν ορισμένες επιχειρήσεις στο κλείσιμο, στο λουκέτο. Άρα η Ισπανική Προεδρία θεώρησε ότι η οδηγία για αυτό το θέμα, τις καθυστερημένες πληρωμές, είναι ε, ύψης της προτεραιότητας. Είναι αναγκαίο το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμφωνήσουν μεταξύ τους οριστικά για αυτό το θέμα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει ακόμα να εγκρίνει, υποφελούμε από αυτή την ευκαιρία, να εγκρίνει εντολή ώστε να ξεκινήσει ο τριμερής διάλογος με την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Εμείς το Συμβούλιο περιμένουμε να προταθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια ημερομηνία για να ξεκινήσει ο τριμερής αυτός διάλογος. Αυτό περιμένουμε. Περιμένουμε να το αποφασίσει αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τη νομοθετική αυτή συζήτηση για την οδηγία που αποτελεί πρόταση προς το παρόν, αλλά δεν πρόκειται για νομική πραγματικότητα ακόμα. έχουμε να κάνουμε με μία περίπλοκη οδηγία, η οποία μάλιστα τεχνικά έχει πολλές και διαφορετικές διαστάσεις. Καλό θα ήταν πάντως να ξεκινήσει ο τριμερής διάλογος όσο γίνεται πιο γρήγορα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχει και ένα τρίτο θέμα, μια τρίτη κατηγορία θεμάτων που έχουν να κάνουν με την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Όσον αφορά αυτό το θέμα, έχουμε διάφορα ζητήματα που εξετάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να ρυθμιστούν. Το θέμα, για παράδειγμα, της πειρατείας, της παραχάραξης. είναι ένα από τα πιο ζημιογόνα φαινόμενα. Ζημιογόνα και για τις καινοτόμες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, αλλά ελοχεύει και κίνδυνος για την ίδια την υγεία των Ευρωπαίων πολιτών. Οπότε το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της 1ης Μαρτίου που μας πέρασε ενέκρινε ψήφισμα βάσει μιας ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου εκφράζει τη θέση του Συμβουλίου για να κερδίσουμε τον αγώνα κατά της πειρατείας και της παραχάραξης. Με ικανοποίηση μπορώ να πω ότι η οδηγία επίσης για θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας έχει ενσωματωθεί στην νομοθεσία όλων των κρατών μελών. Περιμένουμε από την Επιτροπή να μας πει πώς γίνεται στην πράξη εφαρμογή τώρα και πώς προχωράνε τα πράγματα. Έχουμε και τις ε, διατάξεις για τις διαπραγματεύσεις όσον αφορά την παραχάραξη, διαπραγματεύσεις που προχώρησαν πολύ κατά τη διάρκεια του εξαμήνου μας. Και στο θέμα της ε, βιομηχανικής ε, πνευματικής ιδιοκτησίας και τα θέματα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και εδώ είχαμε επαφές με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουμε επίσης προχωρήσει πολύ. Πρέπει να φτάσουμε σε ένα σύστημα κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας για να ενισχύσουμε την ποιότητα της παραγωγής μας, να είναι πιο αποτελεσματικές, ε, πιο σταθερές νομικά οι επιχειρήσεις μας. Πολύ βασικό και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Και θα είναι και ένα όπλο που θα έχει στη διάθεσή της Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσει καλύτερα το διεθνή ανταγωνισμό. Η Ισπανική Προεδρία ελπίζει να βρει μια σωστή, μια καλή λύση και για το γλωσσικό καθεστώς, ώστε να βρεθεί τελικά μια λύση όσον αφορά τα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Θέλω εδώ τέλος να υπογραμμίσω και μια άλλη τέταρτη κατηγορία θεμάτων που έχουν να κάνουν με την εσωτερική αγορά. Πρόκειται για την προστασία των καταναλωτών. Η πρόταση οδηγίας δηλαδή για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Το Συμβούλιο Αγωνιστικότητας, το τελευταίο, της 25ης Μαΐου, συζήτησε επ' αυτού. Νομίζω ότι η συζήτηση ήταν πολύ πλούσια ως προς το περιεχόμενό της, αλλά και πολιτικά ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Υπήρξε σαφής πλειοψηφία υπέρ των θέσεων που στηρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δηλαδή να βρεθεί ένας τρόπος εναρμόνισης μικτός. Και εγώ το στήριξα αυτό εδώ, την προηγούμενη φορά που ήμουνα εδώ μαζί σας. Πέρα δηλαδή από το θέμα της ανώτατης εναρμόνισης, που στην πράξη δεν βοηθούσε και πολύ, πιστεύουμε ότι η νέα θέση του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας θα έχει σαν αποτέλεσμα να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το κείμενο που έχουμε μετά από τη συνάντηση του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας θα το εξετάσει η ομάδα εργασίας στο Συμβούλιο αύριο στις 24 Ιουνίου και είναι πρόταση που έχουμε ετοιμάσει και με τη βελγική κυβέρνηση που αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να καταλήξουμε σε πολιτική συμφωνία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων πριν από τα τέλη της χρονιάς αυτής. Αυτά. Θα ολοκληρώσω αναφερόμενος στον κανονισμό για οι προϊόντα υφαντουργίας. Και εδώ περιμένουμε την εντολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε επί της ουσίας. Έτσι, νομίζω ότι σας μίλησα για όλα τα θέματα τα οποία εξετάσαμε ως Ισπανική Προεδρία για την εσωτερική αγορά. Λίγο πολύ αυτά κάναμε στο Συμβούλιο για τα θέματα που αφορούν την Επιτροπή σας. Τελειώνω, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, υπογραμμίζοντας ότι διανύουμε μία περίοδο κατά την οποία η οικονομική κρίση μας υποχρώνει, και αυτό είναι το θετικό, άμα θέλετε, της οικονομικής κρίσης, να προχωρήσουμε ακόμα πιο γρήγορα προς τα μπρος, να εμβαθύνουμε ακόμα περισσότερο τα θέματα της ενιαίας εσωτερικής αγοράς και τις συνεπιές της. Πιστεύουμε ότι οι κυβερνήσει, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο, η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο, πρέπει να βρεθούν σε ένα κοινό παρονομαστή, ώστε η σημερινή κατάσταση κρίσης να αποτελέσει μια μεγάλη ευκαιρία για πρόοδο και για ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Αναμφίβολα αυτό θα το πετύχουμε με την εσωτερική αγορά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την πολύ πλήρη σας παρουσίαση. Η προσωπική σας δέσμευση για τα θέματα που απασχολούν την Επιτροπή μας είναι πολύ σημαντική. Ε, υπάρχει όντως σημαντική πρόοδος. Διάφοροι ομιλητές θα μιλήσουν τώρα. Η συνάδελφος τώρα θα θέλει να μιλήσει, αύριο θα μιλήσει με τους συντονιστές. Το μόνο άλλο θέμα είναι... Η μόνη άλλη μάλλον είναι η συγγήτρια για... Ε, για τα μέσα με τα οποία θα πετύχουμε την απλούστευση. Είμαστε λίγο απέχουμε. Ε, έχει την εντολή για τη διαπραγμάτευση ε, και δεν έχουμε παραιτηθεί από την ελπίδα να περάσει αυτό το θέμα. Θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους. Ποιος άλλος? Ο Κριστιαν Μπουζόη. Καταρχήν να ευχαριστήσω την ε, Ισπανική Προεδρία. Ήταν πολύ καλή η επικοινωνία αυτών των έξι μηνών μεταξύ Προεδρίας και Κοινοβουλίου. Επίσης, ήταν πολύ καλή η επικοινωνία και με τη δική μας την Επιτροπή και αυτό πολύ σημαντικό. Η εσωτερική αγορά είναι από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομίζω ότι μια καλύτερη οργάνωση και λειτουργία της εσωτερικής αγοράς θα δώσει προστιθέμενη αξία στις προσπάθειές μας καταπολέμησης της κρίσης μεταξύ άλλων. Επίσης θα βοηθήσουμε πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να ξεπεράσουν την κρίση. Μιλήσατε για την έκθεση Μόντι και από ό,τι έχουμε καταλάβει όλοι, πολλά πρέπει ακόμη να γίνουν για την διασφάλιση της καλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Πέρα από την ε, οδηγία για τις υπηρεσίες που είναι πολύ σημαντική για την Επιτροπή μας, υπάρχει και μια άλλη οδηγία που πρέπει να εφαρμοστεί γρήγορα και που εξακολουθεί να έχει κάποια προβλήματα. Πρόκειται για την οδηγία για την επαγγελματική κατάρτιση. Νομίζω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο εδώ. Θέλουμε να εντοπίσουμε αυτή τη στιγμή ποια είναι τα προβλήματα και πώς θα τα ξεπεράσουμε. Έγιναν διαπραγματεύσεις για την μετρολογία, τα κλωστοϊφαντουργικά προϊόντα, για τις, τον τομέα των κατασκευών οικοδομών, στον τομέα των οικοδομών. Αλλά νομίζω ότι επικοδομητικά προσέγγισε τα θέματα αυτά το Συμβούλιο και αυτό είναι καλό. Κάποια στιγμή θα χρειαστεί συμφωνία για τις καθυστερούμενες πληρωμές. Γιατί αυτό είναι από τα μεγαλύτερά μας προβλήματα τώρα και οπωσδήποτε θα βοηθηθούν μέσα από αυτή τη διαδικασία κυρίως οι μικρομεσαίες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι ακόμα Θέλω να σας ε, συγχαρώ για την οδηγία για την διασυνοριακή υγεία, παρόλο που δεν συζητάμε για την υγεία. Είναι από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Ισπανικής Προεδρίας αυτό και ευχαριστούμε άλλη μια φορά. Ευχαριστώ. Μπερνάρ Ζεπανιού, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. Με μικρόφωνο κατά προτίμηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν είμαι στην ίδια πολιτική ομάδα με τον κύριο Μπουσόη, αλλά με πρόλαβε σε κάποια πράγματα. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ισπανική Προεδρία και να τη συγχαρώ πάρα αυτά. Ε, για δύο λόγους. Γιατί, όπως είπε ο κύριος Μπουσόη, ποτέ δεν είχαμε στο παρελθόν τόσο συχνές επαφές ε, με διάφορους υπουργούς ε, της Προεδρίας. Το κάναμε αυτό όμως ε, με την Ισπανική Προεδρία. Εσείς ήρθατε συχνά να μας δείτε για την εσωτερική αγορά, γιατί όπως είπατε η εσωτερική αγορά και η επανέναρξη της όλης διαδικασίας είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά αυτήν την περίοδο. Θέλω να σε ευχαριστήσω, γιατί πραγματικά βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο και βρίσκεστε εσείς στο τιμόνι και νομίζω ότι επειδή ήσασταν η πρώτη προεδρία που ανέλαβε μετά την συνθήκη της Λισαβόνας, τα βρήκατε λίγο μπαστούνια. Έχουμε την προεδρία την κυκλική, δυόμιση χρόνια. Ε, και καταλαβαίνω ότι αντιμετωπίζετε και πολλές ε, εσωτερικές δυσκολίες. Μιλήσατε για την καλή ε, ενσωμάτωση της οδηγίας για τις υπηρεσίες που είναι σημαντικές, σημαντική. Νομίζω ότι έχουμε ήδη προχωρήσει πολύ και στο τέλος του χρόνου θα έχουμε μια καλή αποτίμηση. Ε, τώρα, υπάρχει μια σχέση ανάμεσα στην ε, οδηγία για τις υπηρεσίες και τις επαγγελματικές δεξιότητες, όπως είπε και ο κύριος Μπουσό, Μπουσόη. Είπατε ότι τα αμυγός τομεακά μέτρα δεν αρκούν για να λύσουν την κρίση. Χρειάζονται, μέτρα βιομηχανικής πολιτικής, ε, ε, ευρωπαϊκής έρευνας. Μίλησατε επίσης και για την κατάρτιση αν καταλαβαίνω καλά τόσα λέει ο ισπανικός τύπος, ε, ξεκινήσατε μια μεγάλη πολιτική εκστρατεία για την κατάρτιση των νέων ειδικά, γιατί έχετε και μεγάλη ανεργία στους νέους στη Ισπανία. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτή την ε, ε, προσπάθεια που κάνετε και αυτόν τον προβληματισμό που κάνετε στη Ισπανία τον κάνετε και στην Ευρώπη ε, για τις επαγγελματικές δεξιότητες και προσόντα. Ε, σας ευχαριστώ που ξεκινήσατε αυτή την προσπάθεια. Επίσης, ξεκινήσατε ε, και προχωρήσατε αυτή την οδηγία για την διασυνοριακή περίθαλψη. Ε, πρέπει να προχωρήσει. Θέλω να ευχαριστήσω την Τρινιδά Χιμένες που ε, προωθεί αυτόν τον κανονισμό 883 που εξασφαλίζει μεγαλύτερη ασφάλεια για τους ασθενείς και που είχε σαν σκοπό να εμβαθύνει και να παγιώσει το σύστημα κοινωνικής προστασίας. Για την προστασία των καταναλωτών τέλος, Να ξεκινήσουμε μια πραγματική πολιτική, λοιπόν, όπως ακούσαμε και στην Πάλμα και ελπίζω η Κίνα σιγά σιγά να συνεργαστεί μαζί μας. Πιστεύω ότι όλα αυτά μπορείτε να τα μεταφέρετε στο επόμενο Συμβούλιο, υποβελγική δηλαδή η Προεδρία, που όπως και εσείς έβαλε στο κέντρο της εσωτερικής αγοράς το κοινωνικό χαρακτήρα, γιατί όντως αποτελεί κεντρικό σημείο της. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν και εγώ Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την τελευταία αυτή παρουσίαση στην Επιτροπή μας που ολοκληρώνει μια καλή δουλειά. Μας επιτρέπει να κάνουμε μια ανασκόπηση των πεπραγμένων αλλά και των μη πεπραγμένων. Ε, μετά ε, τη συνθήκη της Λισαβόνας ε, υπήρχαν κάποιες δυσκολίες, δεν είχαμε συνηθίσει, τα κράτη-μέλη κυρίως, ήταν η πρώτη προεδρία μετά. Είχαμε τα, τις καθυστερούμενες πληρωμές, ε, ε, έγινε ακρόαση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτά όλα έδειξαν ότι χρειαζόταν λίγο χρόνος. Ίσως να παίζει ρόλο ο, συγκεκρι... ο συγκεκριμένος φάκελος, ίσως να παίζουν ρόλο οι νέες διαδικασίες μια μικρή ομάδα με τρία μέλη όταν εκπροσωπεί πέντε διαφορετικές απόψεις, εκεί είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Και τέλος, μια δυστυχώς επικριτική παρατήρηση, η αντιμετώπιση του φακέλου late payments, καθυστερούμενες πληρωμές. Θέλαμε μεγαλύτερη συνέπεια, ταχύτερες αντιδράσεις πιο τολμηρές προσεγγίσεις στο θέμα. Θα τα θέλαμε όλα αυτά. Στο Κοινοβούλιο και σε αυτή την Επιτροπή ε, περάσαμε και εμείς από κάποιες αναταράξεις. Καταλήξαμε όμως σε κάποιες συμβιβαστικές λύσεις και περιμέναμε ότι κάτι παρόμοιο θα γινόταν και στο Συμβούλιο. Δυστυχώς όμως δεν έγινε αυτό. Σίγουρα δεν φταίει η Προεδρία η δική σας αλλά ίσως από τους 27 υπάρχουν ακόμα κάποιοι που δεν θέλουν καθόλου να περάσει αυτή η νομοθεσία. Και έτσι, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας, δεν συνεργάστηκαν τόσο επικοδομητικά όσο θα έπρεπε και όπως θα άξιζε ο συγκεκριμένος φάκελος. Ε, σούμα σουμάρουμ λοιπόν από την πλευρά μας εμείς ε, με μεγάλη κατανόηση παρακολουθήσαμε τα θέματα και αν δεν λύθηκε το πρόβλημα των καθυστερούμενων, ε, δεν φταίτε αλλά τα πολλά και διαφορετικά συμφέροντα των 26 κρατών μελών. Ελπίζω όμως ότι αύριο γρήγορα έγκαιρα θα καταλήξουμε σε μία απόφαση. Δεν χρειάζονται πια καθυστερήσεις, γιατί περιμένουν πώς και πώς από εμά οι θυγόμενοι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Μπάρμπαρα Βάιλερ. Και εμείς εκφράζουμε την εκτίμησή μας ως Επιτροπή για το πώς χειρίστηκε το ντοσιέ η κυρία Βάιλερ και ελπίζομαι ότι θα επιτελεστεί πρόοδος πριν τελειώσει ο μήνας. Αυτό είναι προς ε, το καλό όλων. Ο κύριος Τριανταφυλλίδης μετά θα απαντήσει ο κύριος Υπουργός. Ο κύριος Τριανταφυλλίδης. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό για την ε, παρουσίαση του έργου της ε, Προεδρίας θα κάνω τρία-τέσσερα μικρά σχόλια. Σε ό,τι αφορά την προστασία των ε, καταναλωτών, καλωσορίζω την κοινή αντίληψη στην οποία έχει καταλήξει το τελευταίο Συμβούλιο για μειχτή εναρμόνιση. Πιστεύω ότι αυτό βοηθά τις δικές μας συζητήσεις πάνω στο θέμα. Σε ό,τι αφορά την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, έχω την εντύπωση ότι η Ισπανική Προεδρία δεν επεδίωξε την ενίσχυση αυτών των επιχειρήσεων αρκετά. Ε, συγκεντρώθηκε ίσως περισσότερο ε, πάνω στη διάσωση του τραπεζικού συστήματος. Θα ήθελα περισσότερη ε, προσπάθεια σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για την οδηγία για τις υπηρεσίες ήθελα να ρωτήσω πώς αξιολογεί το βαθμό δυσκολίας της μεταφοράς μιας τόσο πολύπλοκης οδηγίας στα νομοθετικά πλαίσια. Ίσως θα πρέπει να δοθεί περισσότερος χρόνος στα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν ε, αυτή την οδηγία για να αποφευθούν προβλήματα. Ε, τέλος, ε, θυμάμαι ότι στην τελευταία επίσκεψη επίσκεψη σας στην Επιτροπή είχατε μιλήσει μέσα στα πλαίσια της του να τονίσετε τη σημασία των διασυνοριακών συναλλαγών και την ανάγκη να ενισχυθεί το διασυνοριακό εμπόριο, αναφερθήκατε στην ε, δημιουργία ενός νέου τύπου ηθαγένειας που να έχει σχέση με την εσωτερική αγορά. Ε, έχουν ληφθεί κάποια μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση και έχει ληφθεί ο παράγοντας καταναλωτής σε αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, ο λόγος στον ε, κύριο Υφυπουργό για να απαντήσει μέχρι τώρα στις ερωτήσεις, στις ερωτήσεις μέχρι τώρα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ, αν μου επιτρέπετε, σε ένα θέμα το οποίο αναφέρθηκε από δύο από εσά. Το θέμα των καθυστερημένων πληρωμών. Και ο κύριος Μπουσόη και η κυρία Πέιλερ αναφέρθηκαν σε αυτό. Η σχετική οδηγία έχει τεράστια σημασία. Και όσον αφορά την υπόθεση πίμες, για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που αναφέρθηκε και ο κύριος Τριανταφυλλίδης για το πόσο μεγάλη σημασία έχουν οι μικρομεσαίες ε, επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ζωτική σημασίας. Και για ορισμένες από αυτές, το θέμα της καθυστέρησης πληρωμών έχει να κάνει με την ίδια τους την ύπαρξη. Σε περίοδο κρίσης, μάλιστα, αποτελεί μία μάστιγα που, μπαίνει, που τις βάζει μάλλον σε ένα φαύλο κύκλο και τις οδηγεί τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε λουκέτο. Εδώ έχει να κάνει και ο δημόσιος τομέας, που και αυτός έχει κάποια ευθύνη, γιατί αν μη τι άλλο θα πρέπει να είναι σε θέση να διορθώσει τις αρνητικές συνέπειες των καθυστερημένων πληρωμών. Μάλιστα, επειδή είμαστε σε μία ενιαία αγορά, υπάρχουν εμπορικές συναλλαγές που είναι υπερεθνικές, διασυνοριακές και άρα το ζήτημα έχει ευρωπαϊκές διαστάσεις είναι ένα ζήτημα που έχει σαν αποτέλεσμα να νομιμοποιείται η ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Γιατί μόνο ευρωπαϊκά μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα των καθυστερημένων πληρωμών σε διασυνοριακές υπερεθνικές συναλλαγές. Σήμερα το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν κάποιες δυσκολίες, όχι όμως επί της ουσίας. Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιες διαφορές όσον αφορά την διαδικασία και υπάρχουν και διαφορές όσον αφορά την ουσία. Και οι μεν και οι δε μπορούν να λυθούν. Όσον αφορά τη διαδικασία, είπα πριν ότι περιμένουμε απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για εντολή προκειμένου να ξεκινήσει ο τριμερής διάλογος. Και με ικανοποιεί ιδιαίτερα η κυρία Πάιλερ με τις καθησυχαστικές της διαβεβαιώσεις. Τώρα από την άλλη υπάρχουν και μερικές διαφορές σε μερικά μόνο σημεία, λίγα, που έχουν να κάνουν με την οδηγία αυτή για την καθυστέρηση πληρωμών. Δεν υπάρχουν ε, διαφορές που να μην μπορέσουν να βρουν λύση ανάμεσα στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σίγουρα θα βρεθεί συνεννόηση. Είναι η χρονική περίοδος για να μπορούν να διαπραγματεύονται τα συμβαλόμενα μέρη. Είναι τα θέματα που έχουν να κάνουν με την υγεία, τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις πληρωμές των δημοσίων αρχών, τα επιτόκια υπερημερίας. Όλα αυτά είναι πράγματα για τα οποία πιστεύω ότι θα βρεθεί κάποια συμφωνία τελικά. Οπότε δεν πιστεύω ότι θα χρειαστεί να μπούμε σε μια μακρά νομοθετική διαδικασία. Εμείς θέλουμε να εγκριθεί συμφωνία πριν τελειώσει η θητεία μας. Αυτή είναι η πρόθεση τουλάχιστον της Ισπανικής Προεδρίας. Λίγες μέρες μας μένουν ακόμα. Θα δουλέψουμε εντατικά λοιπόν, σας διαβεβαιώ, προκειμένου να πετύχουμε την συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν ξεκινήσουν και πάλι οι διαπραγματεύσεις γρήγορα, πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Αναφερθήκατε επίσης, κάποιοι από εσά στο γενικό ζήτημα της εσωτερικής αγοράς. Ο κύριος Μπουσόη και η κυρία Βερνιό αναφέρθηκαν στην εσωτερική αγορά υπό την ευρύτερη έννοια του όρου. Και στις δύο περιπτώσεις από διαφορετική βέβαια οπτική γωνία Αναφερθήκατε στην κατάρτιση των εργαζομένων και των επαγγελματιών. Από τη μία έχουμε τα προσόντα, τα επαγγελματικά προσόντα και από την άλλη μεριά έχουμε την κατάρτιση των νέων. Το τελευταίο αυτό ζήτημα έπαιξε κεντρικό ρόλο στις συζητήσεις μας. Βρίσκεται στο κέντρο εξάλλου της στρατηγικής για το 2020, η κατάρτιση των νέων, η απασχολησιμότητα. Αυτό που ενδιαφέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να υπάρχει κινητικότητα μεταξύ των επαγγελματιών. Άρα η κατάρτιση των επαγγελματιών συνδέεται άμεσα με την κινητικότητά τους. Αυτό είναι προφανές ότι πρέπει να υπάρχει μέσα σε μια νέα αγορά. Οι διάφοροι παράγοντες παραγωγής πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και η παραγωγή να γίνεται εκεί που θα γίνεται πιο αποτελεσματική. Άρα κινητικότητα για να έχουμε την ε, μεγαλύτερη δυνατόν αποτελεσματικότητα. Οι επαγγελματίες πρέπει να μπορούν να βρουν δουλειά εκεί ακριβώς που τους χρειάζονται, εκεί ακριβώς που υπάρχει δουλειά. Οπότε συμφωνώ μαζί σα, κύριε Πουσό και κυρία Βερνιό για τη σημασία που έχει αυτό το θέμα στην εσωτερική αγορά. όλες οι διατυπώσεις για την αναγνώριση των προσόντων πρέπει να προχωρήσουν ακριβώς για να είναι πιο εύκολη η κυκλοφορία των εργαζομένων αλλά και των υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άπαξ ο στόχος για την επόμενη δεκαετία είναι ακριβώς η εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση ως στοιχείο κλειδί για να πετύχουμε την απασχόληση ποιότητα που θέλουμε, άρα και για να είναι βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση ανταγωνιστική, καταλαβαίνετε ότι γι' αυτό του δίνουμε κεντρικό ρόλο. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπορεί να είναι ανταγωνιστική αν πέσουν τα επαγγελματικά προσόντα, αν έχουμε λιγότερης ποιότητας θέσεις απασχόληση, αν πέφτουν οι αμοιβέ. Όχι. Θέλουμε να έχουμε ειδικευμένο προσωπικό με ιδιαίτερα υψηλά προσόντα και γι' αυτό στόχος μας είναι οι νέοι, οι οποίοι απειλούνται περισσότερο. Αφού λοιπόν αυτή είναι η βασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μέλλον, καταλαβαίνετε ότι το θέμα της κινητικότητας των επαγγελματιών, των εργαζομένων, έχει και αυτό κεντρική θέση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς, οι παρατηρήσεις σας είναι παρατηρήσεις που με βρίσκουν πλήρως σύμφωνο. Πολλοί από εσά επίσης και ο κύριος Πουσόη και η κυρία Βερνιό αναφερθήκατε σε ένα από τα πιο σημαντικά νομίζω στοιχεία που πρέπει να υπογραμμίσουμε για την Ισπανική Προεδρία και το Συμβουλίο. Πρόκειται για την διασυνοριακή υγεία. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι γιατί πριν από λίγες μέρες, 7 Ιουνίου όπως γνωρίζετε, το σχετικό συμβούλιο πέτυχε συμφωνία για την οδηγία αυτή. Ήταν μια οδηγία η οποία είχε παραλύσει. Όμως με προσπάθειες προχώρησε. Το ίδιο και για το θέμα για την εγγύηση υπηρεσιών υγείας ποιότητας, αλλά και για την οργάνωση και τη χρηματοδότηση των ε, συστημάτων περίθαλψης των διαφόρων κρατών μελών. Οπότε θέλω να ευχαριστήσω για τα συγχαρητήρια που δώσατε στην Ισπανική Προεδρία για το θέμα αυτό. Όντως και εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντική δουλειά που έχει γίνει από όλα τα θεσμικά όργανα το τελευταίο εξάμεινο. Και για να ολοκληρώσω, θέλω να αναφερθώ στην οδηγία υπηρεσιών. Ο κύριος Μπουσό και, κυρία... και ο κύριος Τριανταφυλλίδης αναφέρθηκαν σε αυτήν και με ρωτήσατε για το πώς προχωράει η εφαρμογή της, πόσο εύκολη δύσκολη είναι η εφαρμογή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάξτε, δεν πιστεύω ότι είναι μια οδηγία ιδιαίτερα εύκολη για να εφαρμοστεί. Όμως είναι αναγκαία, απολύτως αναγκαία. Και επειδή ακριβώ δεν είναι εύκολο να τεθεί σε εφαρμογή γιατί είναι περίπλοκη, νομοθετικά χρειάζονται πολλές μεταρρυθμίσεις σε πολλές χώρες μέλη, γι' αυτό και χρειάζονται παραπάνω προσπάθειες. Η οδηγία για τις υπηρεσίες είναι μια πολύ σημαντική διαρθρωτική μεταρρύθμιση. Σας το είπα και πριν, είναι ζωτική σημασία για την οικονομική ανάκαμψη. Όμως αυτή η οδηγία για τις υπηρεσίες είναι μια οδηγία που απαιτεί ιδιαίτερε προσπάθειες από τα κράτη-μέλη. Εμείς, στην Ισπανία που γνωρίζω και καλύτερα, ολοκληρώσαμε την ε, μεταφορά στην Εθνική Νομοθεσία το 2009 και είμαστε μια χώρα όπου έχουμε μεγάλη αποκέντρωση, όπως ξέρετε. Οπότε δεν είναι μόνο η κεντρική διοίκηση, είναι και οι περιφερειακέ διοικησει και η τοπική αυτοδιοίκηση που πρέπει να θέσουν σε εφαρμογή τώρα αυτή την οδηγία. Είναι αλήθεια, λοιπόν, ότι υπάρχουν δυσκολίες νομικής φύσεως, προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρω και σε όλα τα διοικητικά επίπεδα αυτή η οδηγία. πολύ σημαντικό στοιχείο είναι η διοργανική συνεργασία, η διαθεσμική συνεργασία, η συνεργασία μεταξύ όλων των επιπέδων στις χώρες μέλη ώστε να λειτουργήσει καλά. Δεν φτάνει να εγκριθεί και να εφαρμοστεί από την κεντρική κυβέρνηση η οδηγία αυτή. Αν η τοπική αυτοδιοίκηση, οι περιφερειακές αρχές δεν συνεργαστούν, τότε θα, είναι, θα χωλαίνει η οδηγία αυτή και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα εξακολουθούν να έχουν διοικητικό άχθος, και τη γραφειοκρατία και θα δυσκολεύονται να προχωρήσουν. Συνεπώς, χρειάζεται μέγιστη ελευθέρωση των υπηρεσιών για να είναι πολύ πιο εύκολη η παροχή υπηρεσιών και πιο ανταγωνιστική σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, θα αναφερθώ σε συγκεκριμένα θέματα που μου αναφέρατε. Για παράδειγμα, θα ξεκινήσω με ένα θέμα στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Χάρμπορ στην αρχή. Υπάρχουν ορισμένα θέματα που εκκρεμούν ακόμα, όπως είναι οι πίνακες αντιστοιχίας. Έχουμε προχωρήσει πολύ και θα ολοκληρωθεί το θέμα αυτό υπό Βελγική Προεδρία. Κατά τη διάρκεια δηλαδή που θα είναι οι τρεις προεδρίες μας σε συνεργασία με κοινό πρόγραμμα και άρα με κοινή στρατηγική για 1,5 χρόνο. Ήθελα επίσης να αναφερθώ και σε κάποια πράγματα που είπε η κυρία Βερνιό για την ε, συνεδρίαση στην Πάλμα Ντε Μαγιόρκα. Ήταν ένα σεμινάριο για την ασφάλεια των προϊόντων πριν από μερικές μέρες, 10 και 11 του μηνός. Πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ που πήγατε στο σεμινάριο αυτό. Υπήρξε μεγάλη συμμετοχή από αντιπροσωπείε της Ευρωπαϊκής Ένωση και όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωση, αλλά και από άλλες οικονομίες του ΟΣΑ και είμαι σίγουρο ότι θα μας βοηθήσει η συνάντηση αυτή να προχωρήσουμε και να καταλήξουμε σε συμπεράσματα για να βελτιώσουμε την ασφάλεια των προϊόντων. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς έδειξαν ότι θέλουν να αναθεωρήσουν την Γενική Οδηγία για την Ασφάλεια των Προϊόντων. Θέλουν να βαθύνουν περισσότερο και να συνεργαστούν περισσότερο τελωνιακέ αρχέ, άλλοι φορεί τη αγορά, υπηρεσίε προστασία του καταναλωτή, προκειμένου να έχουν σίγουρα προϊόντα στα χέρια του οι καταναλωτέ. Πολύ σημαντικό και αυτό για να έχει εμπιστοσύνη ο καταναλωτή. Πολύ βασικό αυτό. Νομίζω επίσης ότι η συνάντηση αυτή ήταν μια συνάντηση που κατέδειξε και την εξωτερική διάσταση της εσωτερικής αγοράς. Η έκθεση Μόντι το καταδεικνύει αυτό, ότι υπάρχει αυτή η εξωτερική διάσταση. Δεν πρόκειται μόνο για τις οικονομίες που είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρόκειται και για άλλες οικονομίες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις οποίες έχουμε εμπορικές συναλλαγές. Μπορεί να είμαστε η μεγαλύτερη οικονομική δύναμη του κόσμου, αλλά ακριβώς γι' αυτό η εσωτερική μας αγορά έχει και μια εξωτερική διάσταση. Νομίζω ότι έτσι απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ που εκτιμήσατε θετικά τις προσπάθειες της Ισπανικής Προεδρίας και όχι μόνο της Ισπανικής Προεδρίας όμως. Ε, η αλήθεια είναι ότι μας βοήθησαν πάρα πολύ και οι άλλες 26 χώρες και οι άλλες 26 κυβερνήσεις που συνεργάστηκαν μαζί μας πολύ καλά. Ευχαριστώ λοιπόν για τη συνεργασία και των άλλων θεσμικών οργάνων, γιατί έτσι κι είναι περίπλοκο το Συμβούλιο αλλά ακριβώ γι' αυτό είναι πολύ καλό να έχουμε τη συνεργασία και τη στήριξη των άλλων θεσμικών οργάνων, μεταξύ των οποίων διέπρεψε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Ευχαριστώ για τις δηλώσεις σας, για τις πλήρες απαντήσεις σας. Ε, ακούσαμε την οδηγία για τις πληρωμές. Η κυρία Βάγια θα μιλήσει για αυτή αύριο. Ε, μία σύντομη ερώτηση. Ίσως θα μπορούσατε να μιλήσετε και για το φόρουμ, για την εσωτερική αγορά και τα σχέδια που έχουμε. Φαντάζομαι ότι θα, θα ενδιαφέρεται να εμπλακεί η Ισπανική Προεδρία. Θα μπορούσατε να μας πείτε δύο λόγια για το τι ετοιμάζεται εξ ονόματός μας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Να συγχαρώ και εγώ όπως οι άλλοι συνάδελφοι την Ισπανία για την προεδρία της. Η Ισπανία είναι μία από τις ε, χώρες που βρίσκονται στο προσκήνιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, παίζουν ηθήνοντα ρόλο και βλέπουμε πόσοι πολίτες της Ένωσης ενδιαφέρονται να μάθουν Ισπανικά ε, όχι μόνο επειδή ενδιαφέρονται για τη Λατινική Αμερική, αλλά προπάντων θεωρώ για επειδή ενδιαφέρονται για την Ισπανία. Ε, εύχομαι να ολοκληρωθεί με επιτυχία η Ισπανική Προεδρία ούτω ώστε να εξακολουθεί να συμμετέχει στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών οραμάτων η Ισπανία. Η εσωτερική αγορά ενδείκνυται για την διαμόρφωση και πραγματοποίηση των οραμάτων για την καλύτερη λειτουργία της Ευρώπης. Χαίρομαι που μιλήσατε πολύ για την κινητικότητα, αλλά ακόμα στον τομέα αυτών υπάρχουν πολλά εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν. Η κινητικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τιμωρείται. Δεν μπορούμε τα, τους αριθμούς του τηλεφώνου να τους μεταφέρουμε σε άλλες χώρες. Οι τιμές περιαγωγής εξακολουθούν να είναι πολύ υψηλέ. Ε, πολλά προβλήματα ε, υπάρχουν ακόμη. Όχι μόνο στα πλαίσια των οδηγιών, αλλά και άλλα ζητήματα. Ας δούμε τα δικαιώματα των ταξιδιωτών. Πώς... Ε, εφαρμόζονται στην πράξη. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα μπορέσει να ε, διατηρήσει τον ηθήνοντα ρόλο της Ισπανίας στην Ευρώπη. Είπατε ότι η νομοθεσία δεν φτάνει πάντα στη βάση, στην τοπική αυτοδιοίκηση, για παράδειγμα, στο τοπικό επίπεδο. Ενώ Πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε με τις προσπάθειές μας να φτάσουμε και στο τοπικό επίπεδο, διότι πρώτα θα πρέπει να κοινωνήσουμε τα ενδιαφέροντά μας και βεβαίως θα πρέπει να αρθρώσουν λόγο και οι πολίτες. Γι' αυτό μας ενδιαφέρει στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς να δημιουργήσουμε ένα φόρουμ και ελπίζουμε ότι θα συμμετάσχει και η Ισπανία σε αυτό. Η πρώτη συνεδρίαση θα γίνει επί Βελγικής Προεδρίας και μετά η επόμενη επί Ουγγρικής, αλλά συμμετέχουν όλα τα θεσμικά όργανα. Το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και πολλοί άλλοι ε, εμπλεκόμενοι και θα ήθελα να ανακοινώσω ε, με αυτή την ευκαιρία ότι η πρώτη προπαρασκευαστική συνεδρίαση έγινε και τον Νοέμβριο θα λειτουργήσει το φόρουμ. Ε, ευχαριστώ πολύ. Νόμιζα ότι θα έκανε και ερωτήσει, η κυρία Τούνα. Ε, αν θέλετε να σχολιάσετε, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για την ε, παρέμβασή σας αυτή. Συμφωνώ μαζί σας. με την θετική σας αυτή προσέγγιση όσον αφορά το έργο της Ισπανικής Προεδρίας. Είναι αλήθεια ότι τα ισπανικά είναι μια γλώσσα διεθνής πια. Και είναι μία από τις προσφορές της Ισπανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η γλώσσα μας. Γιατί σίγουρα διευκολύνονται οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με άλλες χώρες στον κόσμο, με, την με τη Λατινική Αμερική για παράδειγμα, που τεράστια περιοχή. Και άρα Πολύ σωστά εκτιμήσατε την προσφορά των Ισπανικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρξε μία συνάντηση το εξάμεινο αυτό στη Μαδρίτη, ε, διάσκεψη κορυφής Ευρωπαϊκή Ένωση Λατινική Αμερική. Ένα από τα πιο θετικά γεγονότα του εξαμήνου αυτού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στραμμένη προς την ε, Λατινική Αμερική. Η Προεδρία μας, δίχως άλλο, είχε κάπως αμερικανική γεύση. Είχαμε τη διάσκεψη αυτή με τη Λατινική Αμερική όπως σας είπα και εκεί είχαμε πολλές ε, συμφωνίες με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Ένα θέμα στο οποίο αναφερθήκατε κι εσείς είναι εκείνο των επιβατών των επιβατών στις αεροπορικές εταιρείες. Ξέρετε ότι φτάνουμε σε μια συμφωνία με τις Ηνωμένε Πολιτείες που ονομάζεται Ανοιχτή Εθέρες, Open Skies. Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Έχει να κάνει και χαίρομαι που το αναφέρατε. Πολύ σωστά. Είναι ζωτική σημασία γιατί πάλι έχουμε να κάνουμε με την κινητικότητα. Η κινητικότητα είναι όρος κλειδί για το παρόν και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όντως, αυτό πρέπει να πετύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση τελικά για όλους τους πολίτες της. Να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα και περισσότερο. Αλλιώς... Είναι σκλαβιά κατά κάποιο τρόπο. Κατά τη γνώμη μου, ο μεγάλος εχθρός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι υπόλοιπα προστατευτισμού υπάρχουν. Και το βλέπουμε αυτό μερικές φορές, ότι υπάρχουν φραγμοί στην κινητικότητα. Η Ευρωπαϊκή Ενία Αγορά συνδέεται άμεσα με τα δικαιώματα των πολιτών. Η Προεδρία μας ήταν μια Προεδρία που συνέπεσε με τη θέση σε ισχύ της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων μαζί με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Η εσωτερική αγορά που συζητάμε εδώ σήμερα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα δικαιώματα των πολιτών και με, με την ευρωπαϊκή ηθαγένεια τώρα τον 21ο αιώνα. Ολοκληρώνω, Πρόεδρε, με το εξή. Χαίρομαι πολύ για την πρωτοβουλία που ελήφθη για το φόρουμ αυτό, η υποβελγική προεδρία. Φυσικά και εμείς θα συμμετάσχουμε. Και δίχως άλλο θα είναι κάτι πολύ χρήσιμο και καινοτόμο. Αποτελεί μία από τις μεγάλες πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μάλιστα, θα λάβει η χώρα η υποβελγικής Προεδρία που συμμετέχει στην τριάδα, στην οποία συμμετέχουμε και εμεί στην τριάδα των προεδρών. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για την ε, δέσμευσή σας, για την επαφή σας με την Επιτροπή μας, ε, για όλα τα θέματα και για τον ενθουσιασμό σας για την εσωτερική αγορά, για την προστασία των καταναλωτών και δύο θέματα που απασχολούν όλο ιδιαίτερο στην Επιτροπή μας. Η δουλειά σας, ε, η υποδοχή της έκθεσης Μόντε και ήταν πολύ σημαντική και η συνέπεια ήταν ο Επίτροπος Μπαρνιέ. Θα προτείνει μια πολύ φιλόδοξη πράξη για την εσωτερική αγορά. Εσείς βοηθήσατε για την κίνηση αυτής της πολύ σημαντικής προσπάθειας. Ε, με μεγάλη χαρά λοιπόν σας υποδεχτήκαμε και σας ακούσαμε. Uh, uh, Κυρίες και κύριοι, και πάμε τώρα στο δεύτερο σημείο της uh, απογευματινής μας ημερήσιας διάταξης, μιας πρώτης δηλαδή ανταλλαγής απόψεων με την εισηγήτρια την κυρία Ευλίν Γκέμπχαρτ για την έκθεση πρωτοβουλίας με σκοπό την εφαρμογή της οδηγίας περί υπηρεσιών. Ακούσαμε, και ήταν καλό αυτό που ακούσαμε από την Ισπανική Προεδρία, τη σημασία που δίνει στην ε, εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Αλλά βεβαίως υπάρχουν πολλά πράγματα που εκκρεμούν που θα τα μελετήσουμε εμείς και που πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν. Θα δώσω το λόγο στην Εύλην. Έχουμε τους σκιώδεις εισηγητές. Δεν ξέρω ποιος είναι ο σκιώδης εισηγητής για τους πράσινους, η Αμελή. Εγώ είμαι σκιώδη εισηγητής για την, το πολιτικό κόμμα το, της Ευρώπης των Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών. Δεν θα σε εκπλήξει αυτό. Κυρία Σβένσον για την ΚΟΕ, δεν είναι εδώ και ο κύριος Σαλίνη Ξέρουμε και το, την τμηματάρχη που εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που θα μας μιλήσει για την εφαρμογή. Εύλην, θα μας μιλήσεις για την έκθεσή σου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για την συνεργασία για μία ακόμη φορά, όχι για το νομοθέτημα, αλλά για να δούμε τώρα πια την πρακτική του εφαρμογή και πώς καταξιώνονται αυτά που ψηφίσαμε στην πράξη. Είχαμε πει ευθύς εξ αρχής στην Επιτροπή ότι οπωσδήποτε θέλαμε ένα νομοθέτημα που δεν θα το ξεχνάγαμε όμως μετά, αλλά θα το ελέγχαμε για να δούμε πώς η νομοθεσία αυτή εφαρμόζεται σε εθνικό επίπεδο και πώς μεταφέρεται στην εθνική νομοθεσία, όχι μόνο στο χαρτί, αλλά και στην πράξη. Είναι σημαντικό το θέμα γιατί είναι ευρύτατη η νομοθεσία και όπως είπε και πριν από λίγο ο κύριος Λόπες πρόκειται για σύνθετη νομοθεσία. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά ήταν και αναγκαία νομοθεσία για να ε, καταφέρουμε δύο τινά. Πρώτον, θέλαμε η αγορά να ανοίξει ε, στις υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πραγματικό άνοιγμα, ούτω ώστε οι άνθρωποι με τις ειδικότητές τους, την εξειδίκευσή τους, τα επαγγέλματά τους, τις δεξιότητές τους να μπορούν να κινούνται ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το δεύτερο είναι ότι η προϋπόθεση θα έπρεπε να είναι η ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών και βεβαίως ε, η ε, διασφάλιση της εφαρμογής του εργατικού δικαίου. Εμείς καταφέραμε να καταλήξουμε σε ένα ισορροπημένο αποτέλεσμα μεταξύ των δύο και γι' αυτό ορίσαμε κάποια σημεία τα οποία ε, πρέπει να ε, εξεταστούν και μέσα από μία μελέτη. Τώρα, μελέτη θα είναι επεξηγηματικό σημείο, μα δεν έχει σημασία πώς θα το πούμε αυτόν τον έλεγχο. Το σημαντικό για μένα είναι το αποτέλεσμα που θα προκύψει από όλα αυτά και που θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Υπάρχει, υπάρχει μια σειρά ερωτήσεων που έπαιξαν ρόλο στην ε, έρευνα αυτή, τη μελέτη αυτή. Είναι αρκετά τα σημαντικά σημεία θεωρώ. Πρώτον, το λεγόμενο screening του ε, εφισταμένου δικαίου και τι νομικές ε, τροποποιήσεις έγιναν στα κράτη-μέλη και πώς λειτουργήσε η νομοθεσία στα κράτη-μέλη. Παραπέμπω πάλι στα λεχθέντα από τον κύριο Λόπες, δηλαδή ότι δεν αρκεί να δούμε τι έγινε σε εθνικό επίπεδο, αλλά σε ομοσπονδιακά κράτη όπως η Ισπανία και η Γερμανία, τι έγινε και το περιφερειακό επίπεδο, στα ομόσπονδα κρατήδια ή στις περιφέρειες της Ισπανίας, για να δώσω αυτά τα δύο παραδείγματα. Πώς δηλαδή η εφαρμογή του screening πραγματοποιήθηκε εκεί. Γιατί η νομοθετική αρμοδιότητα και δικαιοδοσία βρίσκεται σε διαφορετικά επίπεδα. Αλλά νομίζω και στη Γαλλία υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε δηλαδή πώς διαμορφώθηκε στην πράξη η νομοθεσία και πώς λειτουργήσε. Και επίσης ε, και σε άλλα κράτη, από ό,τι αντιλαμβάνουμε υπάρχουν πλέον οριζόντιες και κάθετες διατάξεις, σε ορισμένα μόνο οριζόντιες διατάξεις, σε άλλες χώρες μόνο κάθετες και είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς λειτουργούν όλα αυτά και αν ήταν αρκετά τα μέτρα που ελήφθησαν. Αυτό είναι ένα από τα ερωτήματα που διατυπώνουμε εδώ. Όμως στα πλαίσια του screening ήταν σημαντικό και είναι ένα ακόμα ερώτημα. Δεν θα τα αναφέρω όλα τα ερωτήματα, τις ερωτήσεις. αλλά αναφέρομαι εδώ και σε κάποιες ε, τροπολογίες που πρότειναν οι φιλελεύθεροι και που ευχαρίστως θα τις δεχτώ, δηλαδή να δούμε σε ποιο βαθμό οι παρέχοντες τις ε, υπηρεσίες ε, αλλά και τα συνδικάτα οι οργανώσεις προστασίας καταναλωτών, οι εργοδοτικές οργανώσεις, συμφωνώ να το προσθέσουμε και αυτό. Σε ποιο βαθμό λοιπόν συμπεριλήφθησαν όλοι αυτοί στην αξιολόγηση, γιατί το ευρύτερο αυτό πλαίσιο είναι πολύ σημαντικό εδώ. Το δεύτερο σημείο που θέλω να αναδείξω ιδιαίτερα και δεν θα σας εκπλήξει αυτό βέβαια, είναι οι ενιαίοι εταίροι, ομόλογοι, συνομιλητές αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι το σημαντικότερο μέσον που έχουμε για να λειτουργήσει η οδηγία. Ένα μέσο που επιτρέπει στις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις μικρομεσές, ε, να ε, ωφεληθούν από όλη αυτή την νομοθεσία. Είναι ό,τι πιο χρήσιμο ε, υπάρχει. Με βάση τις πληροφορίες μου Έχω την εντύπωση ότι σε ορισμένα κράτη-μέλη είναι πολύ καλή η κατάσταση. Δεν υπάρχει μόνο μία πύλη στο διαδίκτυο, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι από πίσω, που αυτή ήταν η πρόθεση η αρχική, άνθρωποι που θα βοηθήσουν τις ε, επιχειρήσεις. Και δεν θα είναι μόνο μία πύλη ή μία ιστοσελίδα που θα έχει πληροφορίες μόνο. Δεν επαρκεί αυτό. Και το θέμα των ε, γλωσσών είναι πολύ σημαντικό σε αυτά τα πλαίσια και συμφωνώ κύριε Μπούζο και σε αυτό, δεν ξέρω αν ήταν και ο κύριος Ρόσφορ, ότι θα πρέπει να δούμε δηλαδή σε τι γλώσσες προσφέρονται οι πληροφορίες. Μόνο στη γλώσσα την επίσημη της κάθε ε, χώρας μέλους ή και σε άλλες γλώσσες. Και αυτό είναι σημαντικό. Α, εσείς είσαστε κύριε Λόγκεκάρτ. Δεν θα ήθελα να είναι μόνο αγγλικά, γιατί μπορώ να φανταστώ ότι όταν έχουμε έναν ε, συνομιλητή που είναι στην ε, γαλλική μεθόριο και θα είχε πιο πολύ νόημα να χρησιμοποιηθούν τα γαλλικά και για τα γερμανικά αντίστοιχα στις γερμανικές ή γαλλικές αρχές ε, το ίδιο ισχύει και για τα πολωνικά ή τα αγγλικά, όχι, επουδενή όχι μόνο αγγλικά, ούτω ώστε να έχουμε αυτήν την ε, μονοθυριδική προσέγγιση. Επίσης, το επόμενο που με απασχολεί ιδιαίτερα είναι η διοικητική συνεργασία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, ιδιαίτερα αφού ξέρουμε ότι θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν δυσκολίες μεταξύ διοικήσεων όταν πρόκειται για το δικαίωμα της εγκατάστασης, εξακολουθούν να υφίστανται κανόνες, διατάξεις που πρέπει να ε, εφαρμοστούν, ε, ξουσιοδοτήσεις και σε επαγγέλματα όπου παίζει ρόλο η εξειδίκευση ή κάποιες δεξιότητες συγκεκριμένες να ε, υπάρχει καλή συνεργασία Καλό είναι λοιπόν να συμπεριλάβουμε την πρόταση αυτή για το IMI και να φροντίσουμε να λειτουργήσουν οι προτάσεις. Ίσως όμως θα πρέπει να αναδιατυπώσουμε γιατί στην αρχή δεν κατάλαβα καθόλου τι εννοούσατε. Ίσως ε, ήταν και τόσο περίτεχνα τα αγγλικά σας που εγώ που έχω τα αγγλικά ως τρίτη μου γλώσσα δεν μπορούσα να τα καταλάβω. Πάντως και αυτό το θέμα είναι σημαντικό και θέλουμε να το συμπεριλάβουμε. Επίσης, η αμοιβαία αξιολόγηση. Αυτό είναι σημαντικό θέμα για μένα. Δεν θέλω να το βγάλω, όπως προτείνατε, από, την, το ερωτηματολόγιο. Η αμοιβαία αξιολόγηση αποτελεί μια νεωτερικότητα, ένα, ε, μια καινοτομία που την έχουμε στην ε, οδηγία για τις υπηρεσίες. Σε προηγούμενες οδηγίες δεν υπήρχε αυτό. Οπότε έχει νόημα να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό. Έχει νόημα να ε, ενσωματωθεί αυτό και σε άλλες νομοθεσίες ή είναι περιττό. Για πρώτη φορά έχουμε δημιουργήσει ένα μέσον, ένα μηχανισμό και θέλω να δω λειτουργεί ή δεν λειτουργεί. Παρακαλώ λοιπόν ε, το ΕΛΚ να μην ε, ζητήσει την εξαίρεση αυτού του σημείου από τη μελέτη. Είναι σημαντικό να παραμείνει. Ένα άλλο θέμα που επίσης θα αναφέρω αφορά το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Είναι σημαντικό το πεδίο αυτό και θα πρέπει να, απο... να εξαλείψουμε τυχόν συγχύσεις παρανοήσεις. Δεν πρόκειται μόνο για τις εξαιρέσεις από την οδηγία στην οδηγία για τις υπηρεσίες, αλλά και την οριοθέτηση προς κάθετες οδηγίες που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο το άρθρο 2 αλλά και το άρθρο 3. Προτείνω λοιπόν μια αναδιατύπωση ούτω ώστε να είναι απόλυτα σαφές ότι πρόκειται για το άρθρο 2 και το άρθρο 3 θα πρέπει να καλύπτονται αυτά, ούτω ώστε οι προτάσεις που υπευλήθησαν έχουν σχέση, σύνδεση με την οδηγία αμοιβαίας αναγνώρισης επαγγελματικών τίτλων. Να συμπεριληφθεί και αυτό και ότι όλο το πλαίσιο του άρθρου 3 θα περιλαμβάνεται. Αυτή την ε, επέκταση μπορούμε να την κάνουμε. Αυτά είναι τα θέματα που επέλεξα να παρουσιάσω. Υπάρχουν κι άλλα που μπορεί να μας απασχολήσουν. Αλλά ε, ήθελα να περιοριστώ σε ορισμένα θέματα ώστε να εργαστούμε ταχύτερα. Ε, υποσχέθηκα στον κύριο Σφάμπ στη συνάντηση των ε, συντονιστών να τελειώσει το θέμα και να πάει στην Ολομέλεια το ΔΕΚ. Οπότε δεν μπορεί να είναι τεράστια η μελέτη μας. Αναγκαστικά θα στοχεύσουμε σε συγκεκριμένα σημεία, ώστε να ολοκληρωθεί αυτό το briefing note που το είναι μια έννοια που αντικαθιστά την ε, λέξη μελέτη ε, να έχουμε αυτό το briefing note μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου και πάνω σε αυτή τη βάση να κάνω και εγώ το σχέδιο της έκθεσης και να προβώ στις απαραίτητες προτάσεις. Αυτά είναι τα σημαντικότερα σημεία που ε, θέλω να συμπεριλάβω στο σχέδιο έκθεσής μου. Επίσης, Ε, να σας θυμίσω άλλη μια φορά το χρονοδιάγραμμα όπως το συμφωνήσαμε και στη συνεδρίαση των όπως το συζητήσαμε στη συνεδρίαση των συντονιστών νομίζω ότι είναι εφικτό και θα προβλεφθεί αρκετός χρόνος και για τις τροπολογίες όταν θα κατατεθεί το σχέδιο έκθεσης. Έχουμε σήμερα μια ανταλλαγή απόψεων, μετά τον Ιούλιο, Σεπτέμβριο, σε αυτό το διάστημα θα συναντήσω τους σκιώδεις εισηγητές όλους και βεβαίως θα υποβάλω προτάσεις ε, εκεί για χρονοδιαγράμματα, ούτω ώστε πάνω και στη βάση των ερωτήσεων που έχουμε διαμορφώσει να κάνουμε μια πρώτη συζήτηση και να μου πείτε κι εσείς τι πορεία θα ακολουθήσετε. Μετά θα υπάρξει και ένα workshop εργαστήριο όπου τα briefing notes θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν 29-30 Σεπτεμβρίου μετά εγώ θα καταρτήσω ε, το σχέδιο έκθεσης μέχρι 26-27 Οκτωβρίου θα είναι έτοιμο. 11 Νοεμβρίου θα είναι η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών, οπότε θα έχετε δύο εβδομάδες καιρό περισσότερο από αυτό που προβλέπετε για τις εκθέσεις πρωτοβουλίας, αλλά νομίζω ότι αυτό καλό είναι να το κάνουμε για να γίνει σωστά η δουλειά. Και στις 30 Νοεμβρίου στην ΙΜΚΟ θα ψηφίσουμε, πράγμα που μας επιτρέπει να περάσει στη Σύνοδο του Δεκεμβρίου η έκθεση για να ψηφιστεί εκεί. Είναι σημαντικό να είναι το Δεκέμβριο γιατί στο τέλος του έτους ή στις αρχές του επομένου θα γίνει και η επίσημη αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα κατατεθεί. Οπότε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είμαστε up to date εμείς, για να μην πω ότι θα είμαστε και λίγο ταχύτεροι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, βέβαια μπορεί να, είναι, ε, να συμβαίνει πολλές φορές αυτό, να εργαζόμεθα ταχύτερα. Πάντως, εάν συμπέσουμε ε, στις εργασίες, αυτό πιστεύω ότι θα αναβαθμίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή μας ειδικότερα και είναι και ένα λογικό χρονοδιάγραμμα. Έτσι θα είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες και τα έγγραφα που ήδη έχω λάβει και υποθέτω ότι οι πληροφορίες αυτές θα συνεχίσουν να φτάνουν σε μένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έγκαιρα, ώστε να μπορέσω να δουλέψω πάνω σε σωστή και χρήσιμη βάση. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά προς το παρόν. Ευχαριστώ, Εβελίν, για την πολύ πλήρη παρουσίαση και ελπίζω να συμφωνήσουμε αύριο για τα ενημερωτικά αυτά σημειώματα για να ξεκινήσουμε τη δουλειά, ούτως ώστε να ετοιμαστούμε και να είναι έτοιμη και έκθεση καιρός. Θα δώσω το λόγο σκιώδης κοιόδης από το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι πολύ διότι ξαναρχίζομαι τις εργασίες μας πάνω σε αυτή την οδηγία για τις υπηρεσίες, γιατί θα θυμάστε από την προηγούμενη θητεία ότι ήταν από τα πιο σημαντικά νομοθετήματα και για τους εκπροσώπους των νέων κρατών μελών ε, ήταν πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Αρχίσαμε με αυτό και έπρεπε να θεωρήσαμε ότι είναι ψηλά ο πύχης για μας. Η συνεργασία μας και με την συνάδελφο Γκέμπχαρτ και με τους άλλους συναδέλφους ήταν εξαιρετική και μπορέσαμε να ε, εξετάσουμε το θέμα της εφαρμογής της οδηγίας στα κράτη-μέλη. Τώρα, αν θυμηθούμε τι γινόταν το Δεκέμβριο, ε, θα θυμηθούμε ότι δεν ήταν τόσο ικανοποιητική η κατάσταση στα κράτη-μέλη. Μετά από τους μήνες αυτούς βελτιώθηκαν τα πράγματα, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Είπε ήδη η κυρία Γκέπχαρτ ε, ορισμένα πράγματα για την εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο και το τοπικό επίπεδο. Σε τοπικό επίπεδο Ξέρουν όλοι ότι υπάρχει η οδηγία αυτή ή ακόμα περισσότερο τίθεται το ερώτημα πώς τα κράτη-μέλη θα ενημερώνουν τους επιχειρηματίες για την ύπαρξη της οδηγίας και ότι αυτή την οδηγία μπορούν να την αξιοποιήσουν ή αυτές οι μονοθυριδικές υπηρεσίες ή αν λειτουργεί το σύστημα στην, εθνική, στην επίσημη γλώσσα κάθε χώρας ή και σε άλλες στο Βέλγιο νομοτελειακά θα πρέπει να χρησιμοποιήσω με περισσότερες γλώσσες ενώ στην Πολωνία υπάρχει μόνο η πολωνική γλώσσα ή σε διασυνοριακές συναλλαγές Γερμανία, Πολωνία βέβαια είναι αναγκαστικό να έχουμε και γερμανικά και πολωνικά ε, Επίση από τσέχο-πολωνικά ε, σύνορα θα πρέπει πάλι να υπάρχουν δύο γλώσσες και αυτό ισχύει για όλες τις χώρες και όλα τα σύνορα αν θέλουμε να βοηθήσουμε ε, πραγματικά να βελτιωθούν οι επαφές. Αυτό ήταν ένα από τα ε, ζητήματα τα πιο κέρια στην οδηγία. Επίσης ε, όλοι θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στην διάθεση περισσότερων γλωσσών για την εξυπηρέτηση διασυνοριακών συναλλαγών και επαφών. Επίσης είναι σημαντικό και εμείς οι ευρωβουλευτές πρέπει να το υπογραμμίσουμε αυτό. Νομίζω ότι η έκθεση αυτή θα πρέπει να ασκήσει, αν θέλετε, κάποια πίεση στα κράτη-μέλη, ούτως ώστε να ξέρουν ότι δεν τα αφήνουμε το θέμα να πέσει κάτω. Τι εννοούμε με την άσκηση πιέσεων αν όλοι παρευρισκόμενοι εδώ κάνουμε μια ερώτηση στα κράτη-μέλη σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της οδηγίας, ήδη αυτό αποτελεί μια μορφής πίεση στις κυβερνήσεις μας, στα κράτη-μέλη μας. Τι κάνατε μέχρι τώρα, πώς εφαρμόσατε την οδηγία, πώς την εφαρμόζετε. Ή η διοικητική συνεργασία μεταξύ κρατών μελών υφίσταται αυτό το πράγμα. Λειτουργεί για παράδειγμα, ε, έχουν καταργηθεί όλες οι διατάξεις που είναι ε, ξεπερασμένες. Τι έχει γίνει με τις διοικητικές διαδικασίες. Αυτή η έκθεση λοιπόν θα έχει επίδραση αν και εμείς συμμετέχουμε ε, απευθύνοντας ερωτήματα στις κυβερνήσεις, στους κυβερνητικούς φορείς ζητώντα διευκρινήσεις. Νομίζω ότι η δική μας προσπάθεια θα είναι πολύ σημαντική και θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της έκθεσης. Τέλος θα ήθελα να πω ότι το χρονοδιάγραμμα που προτείνει η Εύλιν Γκέπχαρτ είναι πάρα πολύ ικανοποιητικό και νομίζω ότι μέχρι το Δεκέμβριο θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτό το έργο όλα τα έγγραφα που αναφέρθηκαν θα είναι πολύ χρήσιμα και η πρόταση για τη διοργάνωση του εργαστηρίου, του workshop, είναι πολύ καλή. Γιατί θα δούμε τι θα χρειαστεί να βελτιωθεί, ούτως ώστε να μιλήσουμε για μια σωστή εσωτερική αγορά λειτουργική. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ για την πολύ ενθουσιώδη σας παρουσίαση. Ο κύριος Λουκεγκάρτ που είναι νεοφερμένος στην συζήτηση για την, ε, υπηρεσία, για την οδηγία για τις υπηρεσίες. Καλό είναι να έχουμε και κάποιο φρέσκο πνεύμα, ενώ οι προηγούμενοι ομιλητές ε, είχαν συμμετάσχει στις ε, παλιότερες συζητήσεις όπως και εγώ. Ε, επιτρέψτε μου να μιλήσω δανέζικα, γιατί είναι και νέος το μέσα αυτό. Θα προτιμούσα λοιπόν να μιλήσω τη μητρική μου. Ευχαριστώ. Αυτή η οδηγία είναι η πιο σημαντική οδηγία που έχουμε μπροστά μας, που μας έχει ποτέ απασχολήσει. Όταν σκεφτόμαστε το δυναμικό που έχει αυτή η οδηγία για τις υπηρεσίες, όταν μιλάμε, ε, όταν σκεφτούμε την προσπάθεια καταπολέμησης της κρίσης, το μόνο που θέλω να πω είναι ότι πραγματικά ανυπομονώ να εφαρμοστεί. Γιατί πιστεύω ότι πραγματικά θα πρέπει να στραφούμε και να πιέσουμε τα κράτη-μέλη που δεν έχουν ακόμα κάνει τίποτα. Θα ήθελα όλο το δυναμικό που έχει η αγορά να υλοποιηθεί. Αν εξετάσουμε την έκθεση Μόντι, βλέπουμε ότι ένα πολύ σημαντικό ποσοστό θέσεων απασχόληση εξαρτώνται από αυτήν την οδηγία. Ε, ένα 20% μόνο αποτελούν αντικείμενο διασυνοριακών συναλλαγών. Υπάρχει ένα λοιπόν χαμένο δυναμικό. Είμαστε τώρα σε μια διαδικασία αξιολόγησης. Είναι αυτή η διαδικασία του screening η οποία είναι εξελίξη αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν ακόμα πολλά εμπόδια για να φτάσουμε σε πραγματική εσωτερική ενιαία αγορά. Ορισμένα κρατημέλη δεν έχουν καν εφαρμόσει όλε τι διατάξει. Και αυτό κοστίζει ακριβά. Κάθε μέρα κοστίζει λεφτά αυτό και είναι απαράδεκτο το γεγονό ότι δεν έχει εφαρμοστεί 100%. Ειδικά στα πλαίσια τη κρίση που ζούμε σήμερα. Αυτό που με ανησυχεί πολύ είναι όλα τα κενά, όλες οι ελλείψεις, αυτή η ενιαία μονοαπευθυντική θηρίδα δεν έχει εφαρμοστεί από όλα τα κρατημέλη Μόνο το μισό, το 50% των κρατών μελών έχουν εφαρμόσει αυτή την απέτηση. Τα κράτη-μέλη δίνουν τα δύο τρίτα των πληροφοριών τους στα αγγλικά. Εδώ μιλάμε συνέχεια για τις γλώσσες. Νομίζω ότι στα επιμέρους σύνορα θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερες της μίας γλώσσες. Όταν μιλάμε για τη συνεργασία μεταξύ Πολωνίας και Γερμανίας, ε, είναι ένα πράγμα. Αλλά άλλο αυτή η συνεργασία και άλλο η πανευρωπαϊκή συνεργασία. Όλες οι χώρες εμπλέκονται. Από την άλλη βέβαια υπάρχουν πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που σήμερα δεν τα καταφέρνουν ε, λόγω ε, γλωσσικών φραγμών με αυτή την ενία, στα πλαίσια αυτής της ενίας μόνο απευθυντικής θηρίδας. Ε, Ίσως θα πρέπει να συνοηθούμε ε, πάνω σε μία γλώσσα. Ε, τα αγγλικά, ας πούμε, που λίγο πολύ όλοι τα, τα γνωρίζουμε και τα, και τα μιλάμε. Ε, θα βοηθούσαμε και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αλλά το να επιβάλλουμε 23 διαφορετικές γλώσσες δημιουργούμε ένα απροσπέλαστο τείχος. Σίγουρα θα πρέπει να λύσουμε το γλωσσικό θέμα και τα υπόλοιπα φράγματα, αλλά το γλασικό είναι από τα σημαντικότερα φράγματα. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν. Καταρχάς, η Επιτροπή θα, θα πρέπει να εξακολουθήσει να πιέζει τα κράτη-μέλη, τα οποία δεν έχουν ακόμα μεταφέρει τις διατάξεις της οδηγίας στην εσωτερική τους νομοθεσία. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσει όλους τους μοχλούς πίεσης που έχει στη διάθεσή της για να τα εξαναγκάσει να προχωρήσουν. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε και ένα πίνακα βαθμολόγησης της εσωτερικής αγοράς. Ε, Μέχρι στιγμή ε, τον είχαμε εφαρμόσει αυτόν τον πίνακα και είχαμε επιτυχία. Γιατί όχι και εδώ, στην εσωτερική αγορά. Θα μπορούσαμε λοιπόν να συγκρίνουμε πόσο εφαρμόζει το κάθε κράτο μέλο την οδηγία για την εσωτερική αγορά. Σε άλλου τομεί εφαρμόζουμε αυτόν τον πίνακα βαθμολογία, γιατί όχι και σε αυτόν τον τομέα τη εσωτερική αγορά. Για να μπορούμε να υποδεικνύουμε πούμε, και να στυλιτεύουμε του κακού μαθητέ. Είναι επίση σημαντικό να ενημερώνουμε τι επιχειρήσει γιατί γνωρίζουν πραγματικά τι συμβαίνει. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια έξτρα προσπάθεια ενημέρωσης. Θα πρέπει και οι ίδιε επιχειρήσεις να εμπλακούν στην όλη προσπάθεια. Επίση, στι περιφέρειε, στου Δήμου και στι κοινότητε ε, υπάρχει πλήρη άγνοια ή μια κάποια άγνοια του τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Πρέπει να γίνει μια προσπάθεια ενημέρωση σημαντική. Αυτά ήθελα να σας πω. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Ρούλερ. Θα ήθελα να πω στην προηγούμενη ομιλήτρια ότι στον τομέα της, ε, της οδηγίας των υπηρεσιών έχουν γίνει πολύ περισσότερα πράγματα. Στις 25-26 Μαΐου το Συμβούλιο ασχολήθηκε με την εφαρμογή ε, σε μεγάλες λεπτομέρειες. Αν είχε γίνει αυτό και με άλλες οδηγίες για την οδηγία αυτή για την αμοιβαία αναγνώριση επαγγελματικών δεξιοτήτων θα είχαμε προχωρήσει πολύ. Δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν έγινε τίποτε με την οδηγία των υπηρεσιών, αλλά ένα πρόβλημα είναι ότι είχαμε κάπως υπέρμετρες προσδοκίες. Δεν νομίζω ότι το 60% των υπηρεσιών ε, παρέχονται σε όλη την Ευρώπη. Ε, πολλές είναι σε τοπικό επίπεδο και δεν θα ανοίξουν περισσότερο πανευρωπαϊκά. Ε, εντάξει, να το δεχτούμε αυτό σε ένα βαθμό. Ας μείνει και η εκκλησία στο χωριό, για παράδειγμα. Ε, πάντως, ίσως ε, θα πρέπει να συμμετέχει και η Επιτροπή των Περιφερειών κάποια στιγμή, γιατί η εφαρμογή της οδηγίας ε, κινείται πολύ σε τοπικό περιφερειακό επίπεδο. Οπότε αν ε, διοργανωθεί αυτό το workshop hearing και τι θα είναι, δεν θα ήταν άσχημα να συμμετέχει και η Επιτροπή των Περιφερειών, να προσκληθεί. Ευχαριστώ κυρία Ρούλερ. Ε, και εγώ είμαι σκιώδης ηγητής, να κάνω και εγώ κάποια σχόλια. Το να βασιστούμε στην, ε, βασική, στην καθαρή και ευρύ ενημέρωση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά και αυτό που είπε η κυρία Χάνσεν είναι σημαντικό. Το πώς αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι προ τους απευθύνεται αυτή η οδηγία, την οδηγία αυτή, όπως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έθετε το ερώτημα, έχουμε πετύχει την άρση των διοικητικών φραγμών μέχρι στιγμή και δημιουργούμε νέες ε, επιχειρηματικές ευκαιρίες. Είναι δύσκολο να το απαντήσουμε. Ίσως θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε του φορεί και τι οργανώσει των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να μα βοηθήσουν Στην προσπάθειά μα. Το Eurochambre έχει κάνει μια ανάλυση αναχώρα για τη μεταφορά τη οδηγία στην εσωτερική νομοθεσία στα κράτη-μέλη. Και καλό θα ήταν το Ευρωπαϊκό Επιμελητήριο να μας δώσει αυτές τις πληροφορίες. Ε, νομίζω ότι η μελέτη αυτή ε, δίνει είναι μια προσθέμενη αξία. Δεν ε, αποτελεί επικάλυψη με προηγούμενη δουλειά που έχει γίνει. Επίσης, να ρωτήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν αυτό αυτός ο πίνακα βαθμολογία ε, βοηθάει τι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να παράσχουν διασυνοριακέ υπηρεσίε. Επίσης, από τις ε, πρώτες εμπειρίες που έχουμε από αυτήν την ενιαία θηρίδα, Ε, είναι ενδιαφέρον να μάθουμε τι έχει γίνει. Καλό θα είναι να προσκαλέσουμε τους ε, ανθρώπους που ασχολούνται με αυτά για να μας πούν τι συμβαίνει. Για αυτή την ενιαία θηρίδα. Καλό θα ήταν να ρωτήσουμε πόσο προωθούν τα κράτη-μέλη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, αυτή την ιδέα ότι υπάρχουν νέε ευκαιρίε στην εσωτερική αγορά. Στο Ηνωμένο Βασίλειο με προσκάλεσαν στο πρώτο σεμινάριο που έκανε το, το Υπουργείο Επιχειρήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από έξι μήνε ε, και κάναμε μια συνάντηση με τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Του μιλήσαμε για τι ευκαιρίε που υπάρχουν. Τέτοιου τύπου ε, δραστηριότητε ε, για την υποστήριξη των οργανώσεων επιχειρήσεων είναι σημαντικό. Γιατί πρέπει να μαθαίνουν τι νέε ευκαιρίε που υπάρχουν οι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Θα ήταν κρίμα να μην τι ε, ξέρουν. Η Εύελιν Γκέπχαρτ με ρώτησε με δύο πράγματα για αυτά που είπα για την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνει η κυρία Βαγνιέ και η κυρία Κόμη στην ομάδα προβληματισμού για τα επαγγελματικά προσόντα. Από αυτά που ακούσαμε από κάποιες επαγγελματικές οργανώσεις ε, κατά τη μεταφορά της οδηγίας υπήρχαν ε, θέματα για την ελευθερία παροχής υπηρεσιών διασυνοριακά και πώς αυτό συνδέεται με τις υπάρχουσες ε, προϋποθέσεις για την αμοιβαία αναγνώριση. Μιλάμε για τα επαγγέλματα όπου υπάρχει κινητικότητα. Και εδώ ακριβώς πραγματικά πρέπει να το ψάξουμε για να δούμε αν υπάρχει πρόβλημα. Ε, οι επαγγελματικέ οργάνωση πιστεύουν ότι υπάρχει. Επίση υπάρχουν νέε διατάξει που ανοίγουν ε, την αγορά για τι επαγγελματικέ υπηρεσίε. Παραδείγματο, οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να δημιουργήσουν κοινέ επιχειρήσει. Παραδείγματο χάρη αρχιτέκτονε, ε, δικηγόροι, λογιστές. Είναι πολύ σημαντικό για τα ελεύθερα επαγγέλματα αυτή η δυνατότητα. Και καλό θα ήταν να μα πούνε τι συμβαίνει, πόσε δυνατότητε έχουν να δημιουργήσουν αυτέ τι κοινέ επιχειρήσει. Τελευταίο σχόλιο. Συνδέεται με τη δουλειά που κάνουμε. Νομίζω ότι η δουλειά τη Επιτροπή έχει φτάσει σε ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο, σε μια ενδιαφέρουσα φάση. Ε, εξετάζουμε ε, και αυτή την οδηγία για τι υπηρεσίε και την οδηγία για την αμοιβή αναγνώριση των προσόντων. Ε, όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους Ε, στο τέλος του επόμενου χρόνου ε, θα πρέπει να δούμε πού έχει φτάσει αυτή η οδηγία για την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Ε, επίσης, για τα προσόντα κάναμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση σήμερα το πρωί στην Ακρόαση ε, για την έκθεση Κόζιτσεκ. Παραδείγματο χάρη, ένα εκπρόσωπος του Αυστριακού Εμπορικού Επιμελητήριου ε, είπε ότι σε ορισμένου τομεί υπάρχουν ευρωπαϊκά ε, πρότυπα ποιότητα. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει μία ρήτρα, νομίζω το άρθρο 38, διορθώστε με κάνω λάθο. Υπάρχει, εν στην οδηγία για τι υπηρεσίε ένα άρθρο το οποίο απαιτεί από τα κράτη-μέλη να προωθήσουν ενεργά ε, τα πρότυπα ποιότητα σαν ένα βοήθημα προ του καταναλωτέ. Ε, με την ευρεία έννοια. Μπορεί να είναι και οι επιχειρήσεις, ε, δηλαδή ε, οι συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων ή μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών. Να εθαρίσουν λοιπόν τέτοιου τύπου πρότυπα, ούτως ώστε να βοηθήσουν τους καταναλωτές να κάνουν επιλογές σε άλλες χώρες. Με τη χρήση ευρωπαϊκών λοιπόν προδιαγραφών και προτύπων, ούτω ώστε να ανοίξουν ευκαιρίε γιατί συχνά ε, αποθαρρύνονται ορισμένοι για την παροχή υπηρεσιών ε, διασυνοριακά. Αλλά αν υπήρχαν τέτοιου τύπου προϋποθέσεις, ε, προδιαγραφές, θα διευκολυνόταν αυτή η προσπάθεια. Σε αυτή την έκθεση λοιπόν εφαρμογής θα πρέπει να δούμε πόσο σοβαρά αντιμετωπίζουν αυτή την προϋπόθεση τα κράτη-μέλη. αν υπάρχει πραγματική πρόοδος. Στην έκθεση του εμπορικού επιμελητηρίου δεν υπάρχει τέτοια αναφορά. το ενσωματώνουμε λοιπόν και αυτό στη διαδικασία που είναι να εξελίξει για την οδηγία για τις υπηρεσίες. Ε, περιμένω και προσβλέπω με ανυπομονησία τη συνεργασία με την Εύλην για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα και ελπίζω ότι θα σημειώσουμε και πρόοδο αλλά και θα και θα καταλήξουμε σε σημαντικά πορίσματα, αλλά και κυρίως και πιο σημαντικό σε σημαντικές συστάσεις, ούτως ώστε να είναι αποτελεσματική αυτή η οδηγία. Ε, υπάρχουν και άλλοι ομιλητέ και θέλω να δώσω λόγο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Okay, Mr. Schwab. Ο κύριο Βάμπ είναι ο πρώτο και βεβαίω θα ξαναδώσω το λόγο στην εισηγήτρια για να κλείσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Η Αγγλία προηγείται ένα μηδέν. Σας το λέω αυτό έτσι για να χαλαρώσετε και να ευθυμίσετε. Πέντε σημεία θα προσθέσω. Πρώτον, νομίζω ότι η συζήτηση δείχνει θετικά και νομίζω ότι αναφέρθηκε και από το Σκιώδη ότι οι συζητήσεις που κάναμε το 2006 έχουν ξεπεραστεί, η οδηγία υπάρχει, το είπατε κι εσείς ε, ξεκάθαρα κυρία Γκέπχαρτ, πρέπει να δούμε εάν λειτουργεί σωστά, αν εφαρμόζεται σωστά, που υπάρχουν δυσκολίες. Αυτό πρέπει να κάνουμε τώρα. Δεύτερον, συμφωνώ βέβαια με αυτούς που ασκούν και κάποια κριτική γιατί κάποια κράτη-μέλη καθυστέρησαν αρκετά. Βέβαια, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τη δημιουργία αυτών των μονοθυριδικών υπηρεσιών σε κάποια κράτη-μέλη ε, άλλαξαν άρδιν την διοίκηση ορισμένων κρατών μελών. Βέβαια, καλό είναι να ζητάμε προθυμία, αλλά καλό είναι να δείχνουμε και μια κατανόηση για τις δύσκολες αλλαγές. Αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί προσχηματικά από όλα τα κράτη-μέλη, αλλά γνωρίζουμε τέλος πάντων ότι πρόκειται για μια περίπλοκη διαδικασία, γιατί ε, το ευρωπαϊκό δίκαιο τώρα απαιτεί και μια ευρωπαϊκού τύπου διοίκηση για τα κράτη-μέλη. Να δούμε λοιπόν πώς εφαρμόζουν όλα αυτά τα κράτη-μέλη. Μιλήσατε και για το πεδίο εφαρμογής και η σκιώδης μας η κυρία Χάνσλικ το είπε υπάρχουν πολλά αμφιλεγόμενα θέματα όπου ένας λέει ότι το α άλλο στο β για παράδειγμα οι ε, δάσκαλοι οδήγησης ε, θεωρούν ότι είναι ε, ένας τομέας όπου δεν εφαρμόζεται η οδηγία θα υπάρξουν και άλλα παρόμοια και η ενημέρωση των καταναλωτών είναι σημαντική στο βαθμό που ρυθμίζεται από την οδηγία για τις υπηρεσίες για να δούμε αν είναι ενημερωμένοι όλοι σχετικά με το τι μπορούν να κάνουν με την οδηγία αυτή. Τέταρτον, η εφαρμογή πρέπει να ε, παρακολουθηθεί από τα κράτη-μέλη. Η κυρία Ρούλα έχει δίκιο, αν δούμε δηλαδή τη διαδικασία των συζητήσεων και τη συζητήσει το 2006 βλέπουμε ότι υπάρχει ε, πρόοδος. Θα πρέπει όμως να δούμε και τους ε, επιμέρους κλάδους, να δούμε τι γνώμη έχουν, ποια τα καλά, ποια τα κακά. Το πέμπτο αφορά την αξιολόγηση. Εγώ συμφωνώ με την κυρία Γκέπχαρτ ότι ως κοινοβούλιο θα πρέπει να εξετάσουμε όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται το θέμα, αλλά δεν ξέρω, είμαι λίγο επιφυλακτικός σχετικά με το αν στην έκθεση αυτή πρωτοβουλία έχουμε τη δύναμη να θέσουμε ε, κάποια βασικά θέματα και να καταπιαστούμε με αυτά. Βέβαια μπορούμε να δούμε την αξιολόγηση ε, μέσα από το peer review την αξιολόγηση από ε, ομότιμους φορείς ε, για να δούμε εάν πρόκειται για μια διαδικασία χρήσιμη. Ε, πολύ χαίρομαι που θα συνεργαστούμε και με τη Μάργκοτ και, και με τον Μάλκουλ. Ευχαριστώ, Ανδρέας. Αυτό που είπες συνδέεται με αυτό που είπα και εγώ για την σχέση μεταξύ της οδηγίας για την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και τα επαγγελματικά προσόντα, τα αναγνώριστα των επαγγελματικών προσόντων. Κυρία Βαγνιέ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ προέρχομαι από μια χώρα που δεν υπάρχει αισιοδοξία για την, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της οδηγίας περί υπηρεσιών. Ξεκινήσαμε καθυστερημένα γιατί όταν μιλάμε στη Γαλλία για την οδηγία για υπηρεσίες, μας ε, πηγαίνει το μυαλό στο 2005, ε, διάφορα φαντάσματα ας αρχίζουν να ενσκύπτουν. Υπάρχει κίνδυνο, υπάρχει φόβος. Ε, στη χώρα μου υπήρξε απουσία κοινωνικού διαλόγου. Κάτι που ήταν σημαντικό, όπω είπαν και πολλοί, για την καλή εφαρμογή τη οδηγία. Ορισμένοι είπαν ήταν πολύ σημαντικό για την εσωτερική αγορά και τι θέσει απασχόληση. Υπάρχουν θετικά στοιχεία, αλλά υπάρχουν και αρνητικά. Θα πρέπει να προωθήσουμε τα θετικά στοιχεία. Εγώ έκανα μια μικρή έρευνα στην περιοχή μου στι μικρομεσαίε επιχειρήσει και είπα. Του εξήγησα τι είναι αυτή η οδηγία για τι υπηρεσίε, ε, πώ την ψηφίσαμε, γιατί δεν ξέραν τίποτα, του φόβιζε αυτή η μια θηρίδα τι ήταν αυτό, λέγανε οι επιχειρήσει, ούτε μία δεν τη γνώριζε. Ε, διοικητική συνεργασία. Ξέρετε, οι γαλλικές παραδόσεις τώρα και η γαλλική διοίκηση, η συγκεντρωτική είναι... Έχουμε δυσκολίες να αλλάξουμε. Σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογή, ε, συμφωνώ απόλυτα με την Εύελιν. Ε, έχουμε ένα πρόβλημα με το άρθρο 2 και το άρθρο 3. Προσπαθούμε να το ξαναδούμε, να το δούμε θετικά ε, οι γερουσιαστές μας και η εθνική μας ε, και η Βουλή μας, γιατί υπήρξαν κάποια προβλήματα στην ερμηνεία, κάποιες παρερμηνίες. Αλλά μπορεί να είναι πολύ σημαντικό για τις χιονικές υπηρεσίες, παράδειγμα προς τα μικρά παιδιά και σε μια κρίσιμη περίοδο, σε μια περίοδο κρίσης, όπου η εσωτερική αγορά θα έπρεπε να είναι θετική για κάποιους, αντίθετα ε, δημιουργεί δυσκολίε και μπορεί να στραφεί εναντίον αυτών των ανθρώπων αν υπάρχει κακή εφαρμογή τη οδηγία. Για τα σημεία επαφή, επίση την ενία θηρή θα πρέπει να το ξαναδούμε, ε, με τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Ε, Κάποιο συνάδελφο μίλησε για το ρόλο που μπορεί να παίξει εδώ η Επιτροπή των Περιφερειών. Μέσω τη Επιτροπή των Περιφερειών μπορούμε να προωθήσουμε τα θετικά στοιχεία τη οδηγία ε, στου πολίτε. Ε, να πούμε πού είναι το συμφέρον τους και ποια συμφέροντά τους προωθεί αυτή η οδηγία. Και για το χρονοδιάγραμμα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Συμφωνώ απόλυτα. Ευχαριστώ κυρία Βάγνια. Πρέπει να βρούμε κάποιες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που υποφελούνται από την οδηγία αυτή για τις υπηρεσίες για να δείξουμε τι δυνατότητες επιτυχίας έχει. Η κυρία Τούρινεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ας μιλήσω και εγώ δανέζικα. Περιμένω με ανυπομονησία την, το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας. Πριν εκλεγώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έγιναν μεγάλε συζητήσει, οποίε παρακολούθησα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ήταν στη μέση διάταξη όλων των δανέζικων συζητήσεων. Έγινε μια μεγάλη δημόσια συζήτηση και όλοι για την Ευρωπαϊκή Ένωση μιλούσαν. Δεν θέλω να μιλήσω για την ποιότητα τη συζήτηση, αλλά πάντω έγινε αυτή η συζήτηση στη Δανία. Η δουλειά αυτή είναι πολύ σημαντική. Θα πρέπει να δούμε όλα τα στοιχεία τα οποία μας παρουσίασε η κυρία Γκέπχαρτ, τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα. Υπάρχουν δύο ειδών αξιολογήσεις, μην το ξεχνάμε. Υπάρχει τεχνική αξιολόγηση για να δούμε πώς εφαρμόστηκαν οι διατάξεις ε, της οδηγίας, εφαρμόσαμε τη μονοαπευθυντική θηρίδα. Και υπάρχει και μια πολιτική αξιολόγηση που πρέπει να γίνει οπωσδήποτε. Εξαρτάται βέβαια από την ε, οπτική γωνία. Παραδείγματο χάρη, τι μα απασχολεί, θέσει απασχόληση, σε ποιες συνθήκες ε, δουλεύουμε για τις ε, διασυνοριακές επιχειρήσεις, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, για τις διασυνοριακές υπηρεσίες, συγγνώμη, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τα συνδικάτα. Ο καθένας έχει διαφορετική, ας πούμε, διαφορετικό συμφέρον και ενδιαφέρον. Εγώ σας ευχαριστώ που καλέσατε όλους τους ενδιαφερόμενους σε αυτή την προσπάθεια αξιολόγηση. Είναι σημαντικό να συμμετάσχουν όλοι. Υπάρχει ένα πιο πολιτικό ερώτημα όμως ποια είναι η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται, ποια είναι η εξέλιξη των τιμών, πόσο γίνεται η προσπάθεια, μέσα σε ποιες συνθήκες γίνεται αυτή η προσπάθεια. Εγώ είμαι Δανέζα, που έχει μια καλή σχετικά μπορώ να πω θέση, ε, αγορά εργασίας. Αλλά υπάρχουν και μεγάλες προκλήσεις. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, οι εργαζόμενοι και οι εργάτες περνάνε τα σύνορα υπάρχουν προβλήματα. Δεν νομίζω ότι εφαρμόσαμε όλες τις διατάξεις υπέρ, των εργαζομένων. Δεν μπορούμε να τους πούμε, κοιτάξτε και στο εξωτερικό θα δουλέψετε με τις ίδιες συνθήκες που δουλεύετε στη Δανία. Είναι πολύ σοβαρό αυτό για ένα κοινό project. Θα πρέπει να εξετάσουμε ε, τις συνθήκες εργασίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί οι ευρωπαϊκές οικονομίες βασίζονται όλο και περισσότερο στις υπηρεσίε. Επομένως χρειάζονται ε, αξιοπρεπείς συνθήκε εργασία. Δεν μιλάω μόνο για την Δανία. Είτε Γάλλοι είμαστε, είτε Πολωνοί είμαστε, είτε Δανείοι είμαστε. Θα πρέπει να δουλεύουμε μέσα σε αξιοπρεπεί συνθήκε. Και είναι σημαντικό. Προ το παρόν δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο, στο επιθυμητό επίπεδο. Αυτή είναι η δική μου πολιτική εκτίμηση. Θα πρέπει λοιπόν να καλέσουμε όλου του κοινωνικού εταίρου για να εξετάσουμε σοβαρά αυτό το θέμα. Επίσης είμαι πολύ ικανοποιημένη που θα δουλέψουμε για αυτό το ζήτημα. Ε, συμμετέχω και στην Επιτροπή Απασχόλησης και είμαι σκιώδης εισηγήτρια για τους πράσινους. Θα παρακολουθήσω λοιπόν με μεγάλο ενδιαφέρον την έκθεσή σας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ κυρία Τούρινεν. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που θέλουν να μιλήσουν. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την οποία καλωσορίζω εκ νέου και που παρουσιάζει με μεγάλο ενδιαφέρον ναι, και που παρατηρεί μάλλον μεγάλο ενδιαφέρον την ε, διαδικασία μεταφοράς τη οδηγίες εθνικές νομοθεσίες. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με μεγάλη χαρά επανερχόμαστε στην ε, ΙΜΚΟ για να συζητήσουμε την οδηγία για τις υπηρεσίες. Η Κομισιόν πιστεύει ότι είναι καλή, καλός ο χρονισμός και καλή πρωτοβουλία αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να μας βοηθήσει για να, για να πιέσουμε τα κράτη-μέλη, ούτως ώστε να ολοκληρώσουν τη δουλειά που πρέπει να κάνουν. Η οδηγία για τις υπηρεσίες, όπως υπόθηκε κατ' επανάληψη, και το λέει και ο Επίτροπος Μπαγνιέ συχνά, δεν είναι μια οποιαδήποτε οδηγία, είναι ένα ιδιαίτερο φιλόδοξο πρόγραμμα της ε, ε, εξυγχρονισμού των διοικήσεων των κρατών μελών ε, και το πεδίο εφαρμογή είναι πολύ ευρύ, είναι πολύ μια, μια πολύ δύσκολη προσπάθεια. Τα κράτη-μέλη έκαναν μια καλή προσπάθεια. Βεβαίω υπάρχουν πράγματα ακόμα που δεν έχουν ολοκληρωθεί, πράγματα που πρέπει να γίνουν. Και η Κομισιόν κάνει μια προσπάθεια να εξασφαλίσει ότι θα γίνει αυτή η προσπάθεια. Αυτή την τριετή περίοδο εφαρμογή που δώσαμε στα κράτη-μέλη ήμασταν πολύ δραστήριοι. Αλλά και τώρα που έχει ολοκληρωθεί αυτή η περίοδο, ε, συνεχίζουμε να πιέζουμε με επικοδομητικό τρόπο τα κράτη-μέλη. Ο Επίτροπος Μπαρνιέ το κάνει επίσης ε, σε συνεχείς επαφές που έχει με τις πρωτεύουσε. Ενημερώνουμε και το Συμβούλιο αλλά και το Κοινοβούλιο για την κατάσταση των πραγμάτων σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της οδηγίας. Βλέπετε και τα σημειώματα ε, προς το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας το Μάρτιο και το Μάιο φέτος, ε, ενημερωτικά σημειώματα και Κανένα πρόβλημα δεν είχαμε για να πούμε ποιο κράτος μέλος καθυστερεί κτλ. Θα ήθελα να μιλήσω για κάποιες από τις τεχνικές πτυχές της ε, οδηγίας για την, το σημείο ενιαίας επαφής για τη διοικητική συνεργασία. Έχει συνεχίζεται η δουλειά ε, μέσω του συστήματος ενημέρωσης για την εσωτερική αγορά. Το 2010, φέτος, εξακολουθούμε να πιέζουμε τα κράτη-μέλη για να ολοκληρώσουν την προσπάθειά τους. Ε, και το Κοινοβούλιο από την πλευρά του με τις δικές του εκθέσεις πρωτοβουλίας ε, μας βοηθάει πάρα πολύ. Και εδώ συμφωνώ με τις παρατηρήσεις που έκανε η συγκίτρια κυρία Γκέπχαρτ ότι πρέπει να δράσουμε ταχαίως, στοχευμένα και πρέπει η δουλειά να τελειώσει φέτος. Πρέπει να συνεχιστεί η πίεση. Επίσης, και άλλοι ομιλητές ε, εξέφρασαν την ίδια ευχή να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια. Συμφωνώ. Τι μπορούμε, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη βοήθειά σας. Μπορούμε να πιέσουμε ε, τα κράτη-μέλη για να εφαρμόσουν την νομοθεσία. Η πίεση βοηθάει. Ξέρω ότι διάφορα κράτη-μέλη δεν είχαν ολοκληρώσει την εφαρμογή, αλλά κάθε χρόνο ε, βλέπουμε σε αυτόν τον πίνακα βαθμολογία ότι καθυστερούν τα κράτη-μέλη. Πρέπει λοιπόν ξεκάθαρα να πούμε ότι θα συνεχίσουμε την προσπάθεια, ε, συνεργαζόμαστε. Ε, το Συμβούλιο Δαγωνιστικότητα το Μάρτιο η Κομισιόν έθεσε τις πληροφορίες για τα κράτη-μέλη που καθυστερούν. Τη δεύτερη δεύτερη, στο δεύτερο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας, με το άλλο σημείωμα, ε, είχαμε 8 κράτη-μέλη λιγότερα που, είχαν, ε, που καθυστερούσαν. Χάρη σε αυτή την πίεση, δηλαδή, στο μεσοδιάστημα έγινε αυτή η προσπάθεια. Τώρα για το σημείο ε, ενιαίας επαφής, την ενιαία θηρίδα. Ο κύριος Χάρμπορ είπε ότι θα πρέπει να μας ενημερώσουν ε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η βιομηχανία, οι διάφοροι κλάδοι που θα χρησιμοποιήσουν αυτό το εργαλείο για το πώς πηγαίνει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μία ιδέα που μπορούμε να συζητήσουμε με την εισηγήτρια στις 29 ή 30 Σεπτεμβρίου, αν κατάλαβα καλά, θα οργανώσετε ένα εργαστήρι για να συζητήσετε την έκθεση. Κανονικά στις 30 Σεπτεμβρίου θα γίνει η πρώτη συνάντηση του δικτύου των υπευθύνων για τα σημεία επαφή στα κράτη-μέλη. Αυτό λοιπόν μπορούμε να το συζητήσουμε με την κυρία Κέπχαρτ και με την γραμματεία της ΣΥΜΚΟ όποτε θέλετε. Αλλά αν θέλετε μπορούμε να προσπαθήσουμε οι υπεύθυνοι για τα σημεία επαφή των κρατών μελών να έρθουν εδώ να σας μιλήσουν. Ε, είναι μια ενδιαφέρουσα έτσι, ευκαιρία στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου. Ε, διοικητική συνεργασία, ένα τελευταίο σημείο. Πρέπει και εδώ να πιέσουμε, όχι μόνο ούτως ώστε το σύστημα να λειτουργήσει, αλλά ούτως ώστε οι αρμόδιες αρχές να εξοικειωθούν, να ενημερωθούν για αυτό το θέμα. Η Κομισιόν είναι στη διάθεση της Επιτροπής σας, των, ε, της των σκιωδών εισηγητών, για να σας ενημερώσει, για να σας επικαιροποιήσει τα σημειώματα αυτά τα ενημερωτικά, και περιμένουμε τις ε, μελλοντικές συζητήσεις. Και εγώ σας ευχαριστώ, Κομισιόν, για τη χρήσιμη υπόδειξή σας. Θα δώσω τώρα το λόγο στην εισηγήτρια να κάνει τις καταληκτικές της παρατηρήσεις. Ούτως ή άλλως έχει, μας έχει εξηγήσει ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα. Δεν ξέρω αν θέλει να προσθέσει και κάποια άλλα σημεία. Πάντως περιμένουμε τα συμπεράσματά της. Δεν θα προσθέσω πολλά. Θέλω να ευχαριστήσω τους Κιώδης και τα μέλη που έλαβαν το λόγο. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την εκπεφρασμένη βούληση συνεργασίας για να γίνει το καλύτερο. Όλα αυτά είναι πολύ καλά, επικοδομητικά και αποτελούν καλή βάση για τη δουλειά μας. Θα συνεννοηθώ με τους σκιώδεις για την διοργάνωση του εργαστηρίου. Κατέγραψα τις προτάσεις που έγιναν και μετά θα επεξεργαστούμε εμείς με τη σειρά μας προτάσεις που θα υποβάλλουμε στις, σε μία από τις επόμενες συνεδριάσεις των συντονιστών. Αυτά ήθελα να σας πω και ευχαριστώ. Ευχαριστώ Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Εύλιν Γκέπχαρτ για το εναρκτήριο λάκτισμα. Ευχαριστώ και του όλους όσους παρενέβησαν. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε την συνεδρίαση σήμερα το απόγευμα. Θα επανέλθουμε εδώ, σε αυτή την αίθουσα, αύριο το πρωί στις 9. Και το πρώτο θέμα είναι η έκθεση του Ανδρέα Σβάμπ για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Στις 10 θα αρχίσουν οι ψηφοφορίες. Έχουμε 166 τροπολογίες στην έκθεση αρία, οπότε θα πρέπει να ψηφίσω, Ετσεβερία, συγγνώμη, Αρίας, ε, θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά και γι' αυτό μην ξεχάσετε τι κάρτε σα αύριο. Λοιπόν, διακόπτεται η συνεδρίαση η απόψινή. Τώρα και κλεισμένων των θυρών θα συνεδριάσουν οι συντονιστές.